Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αλλά ε, να ελέγξουμε πρώτα τις ε, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καλώς ήρθατε μετά τις θερινές διακοπές. Ε, τις, ε, ολοκληρώσαμε αισίως ελπίζω και μπορούμε να περάσουμε στις κανονικές μας εργασίες. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά όλους, ε, τα μέλη της Επιτροπής, ε, τη Γραμματεία, τους υπαλλήλους μας, τους διερμηνείς και να περάσουμε στην εξέταση της ημερήσιας διάταξης. Όπως ε, ενημερωθήκατε από τη Γραμματεία, Μία μόνο αλλαγή υπάρχει στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης και αφορά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης με θέμα τις προπτικές και τις ευκαιρίες ε, της ευρωπαϊκής ε, μελισσοκομείας. Αναβάλλεται για αύριο στις 9 η παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Ως εκ τούτου η παρουσίαση του ΣΤΟΑ για την γεωργία ακριβίας και το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα ως σημείο 11. εξηγητή τη σχετική έκθεση είναι ο κύριο Ερντό. Ελπίζω να γίνει δεκτή η ημερήσια διάταξη. Με την αλλαγή αυτή ευχαριστώ. Έχουμε απευθεία αναμετάδοση από το διαδίκτυο τη συνεδρίασης και ε, διερμηνία έχουμε σε 20 γλώσσε με εξαίρεση τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κερτικά, κοεδελικά. Σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 12 Ιουνίου και 19 20 Ιουνίου, ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία. Και περνάμε στο σημείο 4, το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοσιονομική Χρήση 2018. Όλα τα τμήματα. Ε, η συγητής μας είναι ο κύριος Τίμπορ Σάνι. Είχαμε ήδη ακούσει την παρουσίαση την προηγούμενη φορά. και στις 11 Ιουλίου μας παρουσίασε το σχέδιο γραμματότησής του με ε, συγκεκριμένα κονδύλια που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο και πάλι ο εισηγητής μας, ο κύριος Σάνι. Παρακαλώ αν έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που μας είχατε πει την περασμένη φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ όλους σας μετά τις ε, ωραίες αυτές α, θερινές διακοπές. Θα είμαι σύντομος όπως μου ζητήσατε. Ε, δυστυχώς ε, το εξαιρετικό καλοκαίρι δεν ε, ήταν ευνοϊκό για έντονες διαπραγματεύσεις. Πάντως μετά τις τελευταίες δύο μέρες όπου επανήλθαμε όλοι οι συνάδελφοι έδειξαν πολύ μεγάλη προσήλωση στο θέμα και ευχαριστώ θερ, θερμά την Κατερίνα, τον και για την πολύτιμη βοήθειά τους και μας βοήθησαν να περάσουμε στην τελική ευθεία αυτού του θέματος. Νομίζω ότι μπορούμε πια να συμπεριλάβουμε σχεδόν όλα τα σχόλια και τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων και θεωρώ ότι η έκθεση μου τώρα περιλαμβάνει όλες τις ε, σημαντικές θέσεις μας ε, του τελευταίου εξαμήνου έως και χρόνου. Είναι πολύ θετικό ο κατάλογος ψηφοφορίας, είδατε ότι βρήθη θετικών προσήμων, οπότε ελπίζω αυτή την, ε, αυτό το θετικό πνεύμα να πρετανεύσει και στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Ωραία, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία του κυρίου Βιέγκας. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Εγκρίνεται.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 Mamy przegłosować jeszcze poprawkę. Θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία 3. Επιστρέφουμε στην 3. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Και τώρα την 6 Τροπολογία 6. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 1. Τέλο ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παίρνουμε στην τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 16. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 του κυρίου Βούδα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 τον Καπούτο και Σάνι. Ποιος είναι υπέρ της 49. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 51 του κυρίου Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 52 της κυρίας Ένερα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 52. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τροπολογία 30 τον Γιάρ και Μαγκίνες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. επανάληψη της ψηφοφορίας, γιατί βιάστηκα λίγο, επανάληψη της ψηφοφορίας του σχεδίου γνωμοδότης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Προλάβετε να ψηφίσετε τώρα. Ωραία, οπότε λίγη ψηφοφορία. Ευχαριστώ που με επισημάνατε αυτή τη βιασύνη εγκρίνεται και περνάμε στο σημείο 5 την έκθεση της αρμόδιας καθήλη επιτροπής και πάλι η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Τίμπορ Σάνι καλύτερα να του δώσω λοιπόν το λόγο για να μας κατατοπίσει ή μήπως δεν θέλετε δεν θέλετε οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία Τροπολογία 62-37. Ε, θα λέω μόνο το τελευταίο σημείο. Ποιος είναι υπέρ τη 62-37. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 62-38. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 69. 39, συγγνώμη. 62-39. Εγκρίνεται. 62-40. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 41 υπέρ εγκρίνεται. 42. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 43. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 45 υπέρ εγκρίνεται 34 υπέρ εγκρίνεται 12 υπέρ εγκρίνεται 15 υπέρ εγκρίνεται Η 15 καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκε η 62-12. 62-16, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62-07 του κυρίου Γιάρ, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 6209 του κυρίου Γιάρη Περ εγκρίνεται. Η τροπολογία που λύγει σε 20. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η τροπολογία που λύγει σε 11. Υπέρ. Εγκρίνεται. 62-11 λέει πάλι υπερ Υπέρ, εγκρίνεται. 62-06, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 62-08, υπέρ, εγκρίνεται. 62-14, τα κούλα και άλλων, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62-21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-22. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 47. Του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 62-10. και 62-13 πανομοιότυπες. Ψηφίζουμε μαζί υπέρ, εγκρίνονται. 14 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 48 υπέρ, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 25. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά, οπότε καλώς τα ελέγξαμε. Δεν φαινόταν ε, με το μάτι. 32 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 50 υπέρ, εγκρίνεται. Ο εισηγητή δεν ψηφίζει τις δικές του τροπολογίες, βλέπω. Τροπολογία 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Εγκρίνεται. 62 62.00. Κυρίων Σάνι και Μπόκοβιτς. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 62.03. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται με μικρή διαφορά εξού και η εξακρίβωση 62.04 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται τροπολογία Ανδρία και 05 υπέρ κατά Απορρίπτεται, τέλο στο ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 6205. Τέλο ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6218. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 30, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 57 του εισηγητού, ποιος είναι υπέρ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 6202. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. «58 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 του εισηγητού. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 του εισηγητού. Υπέρ. Εγκρίνεται. 61 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 64 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 65 υπέρ εγκρίνεται. 66 υπέρ εγκρίνεται. 62-01 ε, συγγνώμη υπέρ εγκρίνεται. συγγνώμη, ξέχασα την 62-67. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 62-19, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την ψηφοφορία για το σημείο 5 και περνάμε στο σημείο 6. Σας ευχαριστώ καταφέραμε και διεκπαιρεώσαμε αισίως την ψηφοφορία και ευχαριστώ τον εισηγητή για τις δύο γνωμοδοτήσεις του. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Ο κύριο Σάνι. Έχετε το λόγο κύριε Σάνι, αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να πω κάτι πολύ συμβολικό. Νο πασαράν, δεν θα περάσουν. Ευχαριστώ και περνάω στο σημείο 6. Η προσαρμογή ευθυγράμμιση νομικών πράξεων ε, που προβλέπουν ε, τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας ε, με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριτής είναι ο κύριος Ντάνιελ Μπούντα, συγκεκριτή γνωμοδότησης και αρμόδιος για την σύνταξη της έκθεσης στην αρμόδια καθήλη επιτροπή είναι ο κύριος Σάιερ. Καλύτερα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπούντα, για να μην σας καθυστερώ εγώ, να μας την παρουσιάσει ο κύριος Μπούντα και να ψηφίσουμε. Δεν θέλει το λόγο όμως ο εισηγητής ο κύριος Μπούντα, οπότε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Προτείνουμε μάλιστα να ψηφίζουμε ομαδών τις τροπολογίες, γιατί πολλές τροπολογίες 197 είναι συνολικά, αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία μαζί όλων των τροπολογιών, που είναι κυρίως του κυρίου Καπούτο και άλλων βέβαια, αλλά η πλειοψηφία των πλειονότητα των τροπολογιών του κυρίου Καπούτο. Άρχεται η ψηφοφορία συνολικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται 197 τροπολογίες του κυρίου Καπούτο. Περνάμε στις υπόλοιπες τώρα. Τροπολογία 7 του κυρίου Ερντός. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 7 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91 και 92. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 148. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 149 και τροπολογία 150. Από ταυτόσημες υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογίες 151 και 152 παρόμοιε υπέρ. Εγκρίνονται. 157. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται 158 υπέρ κατά απορρίπτεται 159 υπέρ κατά απορρίπτεται 160 υπέρ κατά απορρίπτεται 161, 162, 163 παρόμοιε υπέρ εγκρίνονται 164, 165 Ποιο είναι υπέρ εγκρίνονται 166 υπέρ κατά απορρίπτεται 168 Ποιο είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 169 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολόγες 1, 170 και 171 ταυτόσημες, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. 178 του κυρίου Νέκοφ, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά απορρίπτεται. 182 και 183 παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 191 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 195 και 166 υπέρ, εγκρίνονται. 198 δεν ψηφίζουμε γιατί είναι τεχνική φύσεως. 199 το ίδιο. Πάμε στη 200. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2. Μάλλον εγκρίνεται. Αλλά επειδή σηκώσετε το χέρι όλοι, Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η αριστερή πλευρά της αίθουσας δεν ψήφισε. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να διαπιστώσω το αποτέλεσμα. Αλλά όπως σας είπα ήμουν βέβαιος ότι είχε εγκριθεί η τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 202 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, 202 του κ. Φλάναγκα, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Τροπολογίες 5 και 204. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνονται. 205 και 206 παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 6 του κυρίου Αρντός. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης μετά την έγκριση των τροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κύριου Μπούντα. Δεν ξέρω αν ο συγγετής μας θέλει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους στη γνωμοδότηση αυτή. Προσωπικά, πρέπει να σας πω ότι έλαβα υπόψη μου και τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στις κατεξουδότησης πράξης. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Όντω ήταν σημαντική αυτή η γνωμοδότηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μας και μπορούμε να περάσουμε στις συζητήσεις επί της ουσίας για τα υπόλοιπα σημεία. Πρώτα, σημείο 7, συστάσεις για τη διαπραγματευτική εντολή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία εισηγητής της ε, Γνωμοδότηση είναι ο κύριο Αντριέ. Πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση, γιατί γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι η θέση της Αυστραλίας στις παγκόσμιες γεωρικές αγορές και πόσο θα επηρεάσει τις εμπορικές μας σχέσεις ε, μια τέτοια συμφωνία και κυρίως τη Γεωργία. θέλουμε να αναλυθεί υπόψη η θέση Ευρωπαϊκής, ε, της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό προβλέψαμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να μπορέσει η αρμόδια για το Διεθνές Εμπόριο Επιτροπή και κατόπιν η Ολομέλεια να επιληφθούν σε σχετικά σύντομο διάστημα ώστε το ψήφισμα να το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς, ε, επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός διαδικασίας, δεν μπορέσετε να καταθέσετε τροπολογίες με βάση το σύστημα AT4AM, αλλά οι Γραμματεία ενημέρωση πώ μπορείτε χρησιμοποιώντα έγγραφο Word να υποβάλλετε ψηφοφορίε που έπρεπε να τι στείλετε στη γραμματεία μέχρι την 1η Ενάτου στι 11 το μεσημέρι. Δύο μέρε ακόμη λοιπόν για να λήξει η διορία για την υποβολή τροπολογιών. Ο κύριο Ανδρέα απουσιάζει, οπότε δεν μπορεί να σα παρουσιάσει προσωπικά την γνωμοδότησή του. Ο κύριος Δενανό όμως θα τον αντικαταστήσει και θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση του κυρίου Αντρία. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Δενανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ο Ρικ Αντριέ δεν ε, ε, μπορεί να παρευρίσκεται γιατί έχει ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Θα σας αναγνώσω εγώ το σχέδιο νομοδότησης του. Λέει ότι η γεωργία χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το πιο ευαίσθητο τμήμα αυτού του σχεδίου συμφωνίας. Η ε, Αυστραλία έχει μια μεγάλη γκάμα παραγωγή γεωργικών προϊόντων, κυρίως για την εξαγωγή. Μετά τη Βραζιλία και την Ελλάδα είναι η τρίτη ε, εξαγωγική χώρα στη ζάχαρη και επίσης έχει πολύ μεγάλη κτηνοτροφία με πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες κτηνοτροφίας. 60% των βοηδών και των ε, εγωπροβάτων ε, απευθύνονται, μάλλον προορίζονται για τις εξαγωγές, όπως και η Βραζιλία. Το 1986 στον κύριο της Ουρουγουάης ε, ήταν ιδρυτικό μέλος ε, των εξαγωγικών χωρών. Ήδη χρησιμοποιεί όλες τις ποσοστώσεις που ε, διαθέτει και την ευνοούν. Έχει ως απαιτήσει την άρση των δασμολογικών φραγμών. Θα έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα ε, αν ανοίξει η αγορά σε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενώ ε, αντίστροφα είναι περιορισμένο το δικό μας ενδιαφέρον γιατί είναι μόλις 23 εκατομμύρια οι Αυστραλοί. Άρα ε, θέλω να προχωρήσω σε συστάσεις και προειδοποιήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής μας, λέει ο κύριος Αντριού. Θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε είδους ανισορροπία ε, εις βάρος γεωργίας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν θα πρέπει και πάλι να είναι το τίμημα, Γεωργία, το αντάλλαγμα για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση ε, στην ε, αγορά της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες και τα βιομηχανικά προϊόντα. Ε, το πρόβιο κρέας, το βόλιο κρέας, τα δημητριακά και η ζάχαρη θα πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηριστούν ευαίσθητοι τομεί. Γιατί είναι πάρα πολύ εύθραυστες αυτές οι συμφωνίες με την Αυστραλία και για τομείς όπως είναι ε, ε, ζάχαρη από ειδικά προϊόντα που αφορούν τις δικές μας υπερπόντιες ε, περιφέρειες και το βόλιο και το πρόβιο κρέας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλες τις αποστώσεις και τις ειδικέ ευνοϊκές συνθήκες που έχει η Αυστραλία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης και τις επιπτώσεις του Brexit και πώς μπορούμε ακόμα να κάνουμε παραχωρήσεις προς την Αυστραλία. Αν παραμείνουμε σε αυτή τη γραμμή, δεν θα πρέπει να ποντάρουμε μόνο στους δασμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει τη μάχη για άλλα εμπόδια, άλλους φραγμούς τεχνικούς, υγειονομικούς, αλλά και δείξεις γεωγραφικής προέλευσης αν δεν ληφθούν αυτά υπόψη, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συμφωνία. Αυτά σας διάβασα, αυτά που λέει ο κύριος Ανατολή και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Περάμε στη συζήτηση. Παρακαλώ να μην μακρηγορείτε. Κυρία Μίλλερ. Κυρία Μίλλερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, θα ήθελα κι εγώ εξ ονόματος του συναδέλφου Τάκουλα να παρουσιάσω τη δική μας νομοδότηση. Συχώς κολλείεται και ο κύριος Τάκουλα και μου έδωσε ένα χαρτί με μερικά σημεία να διαβάσω. Η Ευρώπη χρειάζεται μια φιλόδοξη, ε, ευρύτερη, ε, συνολική συμφωνία με ε, την Αυστραλία που να λαμβάνει υπόψη ευαίσθητους και ε, κρίσιμους τομείς όπως είναι το γάλα, το ε, βόηο, το πρόβιο κρέας κτλ. Θα πρέπει να έχουν ευκαιρία όλοι οι παραγωγοί και οι Ευρωπαίοι και οι Αυστραλοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος παγκοσμίω, θα πρέπει να προωθούμε τη θέση αυτή και πρόκειται να αρχίσουμε μια διαπραγμάτευση με ένα μεγάλο παραγωγό γεωργικών προϊόντων και είστε θέμα και ανταγωνιστικότητα τη δική μας γεωργίας. Ο εισηγητή έχει μια γραμμή, να συντάξει καλύτερα της νομοδότηση, που είναι για μας υπερβολικά κριτική. Θα κάνουμε τροπολογίες, δεν τα βλέπουμε τόσο αρνητικά δεν μπορούμε να θεωρούμε αποκλειστικά απειλή την ε, αγορά γεωργικών προϊόντων της Αυστραλίας. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη χώρα και ξέρω τι τραβάει από τη λειψιδρία, την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή γενικότερα. Υπάρχουν περιφέρειες όπου η παραγωγή είναι πολύ καλή και πολύ εύκολη, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες. Άρα θα πρέπει εμείς προφανώς να είμαστε στο πλευρό ε, της ευρωπαϊκής γεωργικής αγοράς με απαιτήσει, αλλά να σκεφτούμε ε, που θα ζητήσουμε ποσοστώσεις και ποιες. Βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ευαίσθητοι τομείς και χρειάζεται εκεί διαπραγμάτευση. Υπάρχει και δυνατότητα για διαπραγμάτευση και για προστασία μας. Παρόλα αυτά παραμένουμε ε, θετικά διακείμενη για την εμπορική αυτή συμφωνία, για την ευκαιρία όχι μόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για την ευρωπαϊκή γεωργία ανοίγεται ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Εάν είμαστε μεθοδικοί και συστηματικοί στη δουλειά μας μπορούμε να έχουμε την ε, Αυστραλία ως ισότιμο εταίρο ε, και εμπορικό για να τη δεχτούμε και να κάνουμε και δουλειές και να συνεργαστούμε με τους Αυστραλούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκολσον. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ εισηγητή για τη γνωμοδότηση για τη Νέα Ζηλανδία και θα μιλήσω στο επόμενο. Επομένω, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων εάν ε, επαναλάβω τα ίδια πράγματα, διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία, η οποία θα μπορέσει να προσφέρει πάρα πολλέ ευκαιρίε, εάν μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συμφωνία. Υπάρχουν ευαίσθητοι τομεί ε, ε, για τον τομέα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, τους οποίους πρέπει να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε. Οι τελικές συνέπειες εκχωρήσεων στην ε, γεωργία σε συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, συναυτοί, θα πρέπει να λεφθούν υπόψη. Και επίσης πρέπει να δούμε τι πιθανά κέρδη και απώλειες μπορεί να έχουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί με αυτή τη μελλοντική συμφωνία. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκπώνησε και μία μελέτη για το ε, τι ε, τρόφιμα θα μπορούσε να καταναλώσει η Ευρώπη ενεργά μέσω αυτών των συμφωνιών. Δεν έχω ακούσει όμως ε, κάτι τελικά για την έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πού υπάρχει στήριξη, τι περιλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση αν υπάρχει, ε, πριν προχωρήσουμε στις επόμενες εμπορικές συμφωνίες. Δεν είμαι κατά των συμφωνιών, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς ε, περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Μου τα είχε πει ο κύριος Χόγκαν, αν θυμάμαι καλά, και θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσον εξετάστηκαν. Ε, Βέβαια, υπάρχουν εξαιρετικέ δυνατότητε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή τη συμφωνία. Η Αυστραλία είναι 24 εκατομμύρια άνθρωποι και επομένω ε, ε, υπάρχουν και πολύ σημαντικέ σχέσει. Το 2016 υπήρχε διμερές ε, εμπόριο γεωργίας ε, μεγάλου κύκλου εργασιών. Και επίσης θα πρέπει να δω και το σημείο 7 του σχεδίου έκθεσης που αφορά το Brexit. Ξέρουμε ότι το Brexit θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς Γεωργίας. Αλλά εγώ ως μέλος ανησυχώ αν λέμε στους άλλους 27 τι να κάνουν και να χρησιμοποιείτε το Brexit ως δικαιολογία ε, για το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται σε θέματα εμπορίου. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί απάντηση αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Oui, merci, monsieur Président. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τις ε, προτάσεις του κειμένου, πέραν του σημείου 8, ε, δεν έχουμε κάτι ευνοϊκό για το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Δείχνουν πόσο πολύ ευάλωτο είναι ο γεωργικό τομέα ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι τέτοιες συμφωνίες θα ήταν καταστροφικές, για τον τομέα μα. Ε, μετά τη Βραζιλία υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα στη θέματα κτηνοτροφίας. Να υπενθυμίσω ότι το 60% του κρέατος που εξάγεται είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ποσοστό. Πρέπει να ε, αποκλειστεί το βόηο κρέας και το κρέας των πουλερικών όπως προτείνεται στο σημείο 5 και να υπάρχουν εμπορικές σχέσεις σε τομείς στους οποίους δεν υπάρχει ανταγωνισμός θα πρέπει να αφήσουμε τη δυνατότητα κάθε κυρίαρχη χώρα να διαπραγματευτεί μόνη τη μια συμφωνία και να μην υποστούμε ε, στη συνέχεια τέτοιες αυτοκτονικές ε, συμφωνίε. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη ε, διότι εγώ επισκέπτομαι ως ε, μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και πολύ στενά τα θέματα, παρακολουθώ τα θέματα αυτά και πίστευα ότι θα ήταν καλό να ακούσω ε, εδώ απευθείας τι συζητάτε στην Επιτροπή σας για το θέμα αυτό. Διαβάζοντας τα κείμενα ε, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν αντανακλώνται συνήθως αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοι και θεώρησα λοιπόν ότι είναι καλή ευκαιρία να έρθω εδώ να τα ακούσω αυτά διαζώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια ανοιχτή αγροδιατροφική αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τομέα της γεωργίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ε, γεωργικών ε, διατροφικών προϊόντων. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι εύκολα και ότι ε, το θέμα αυτό είναι εύκολα. Ε, το βόλιο κρέας αναφέρθηκε από αρκετούς συναδέλφους, είναι αρκετά ευαίσθητος τομέας, υπάρχουν αρκετές ευαισθησίες στον τομέα αυτό. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η αγωγή βόηου κρέας από την Αυστραλία είναι 24 εκατομμύρια τόνοι και καταναλώνται 8 8 ε, εκατομμύρια τόνοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ποσοστό αυτό. Ξεκινάμε από πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο ε, στην Αυστραλία. Ελπίζω λοιπόν να ακούσω και κάποιες ε, σκέψεις σας και κάπου στο ε, οριστικό κείμενο να υπάρχουν και κάποια ε, επιθετικά συμφέροντα. Ξέρετε ότι υπάρχουν και επιθετικά συμφέροντα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο εμπόριο με την Αυστραλία. Και ένα από τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε σαφέστατα αυτή τη στιγμή είναι ότι μα ενδιαφέρει το τυρί το οποίο εξάγεται αυτή τη στιγμή. Ε, 154 εκατομμύρια ευρώ είναι ο κύκλο εργασιών και εισάγεται μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ ε, ε σε ποσότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά και επιθετικά συμφέροντα και φυσικά και αρκετά λεπτά ζητήματα και συμφέροντα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Παραδείγματο χάρη κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμένα είναι η εξαγωγή ίνου. Στην Αυστραλία η αγορά του ίνου είναι ε, αρκετά ε, Ζαθροί, υπάρχουν προβλήματα. Εμείς είμαστε καθαρή εισαγωγή ε, ε, ε, ίνου από την Αυστραλία. 136 εκατομμύρια αξίας ίνου έχουμε και εξάγονται μόνο 88 εκατομμύρια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν είναι Πώ είναι δυνατόν αυτό, γνωρίζοντα ότι τα ευρωπαϊκά κρασιά είναι παγκοσμίω γνωστά ως τα καλύτερα στον κόσμο. Εάν ε, λοιπόν ψάξουμε το θέμα λίγο παραπάνω, θα δούμε ότι υπάρχουν υψηλοί δασμοί στην Αυστραλία για τα ευρωπαϊκά κρασιά και υπάρχει και ένα πολύ ε, αυστηρό σύστημα εισαγωγών για το ευρωπαϊκό κρασί. Επομένως υπάρχουν κάποιοι τομείς τους οποίους πρέπει να εξετάσουμε λίγο καλύτερα και ελπίζω να μπορέσετε κι εσείς να συμβάλλετε από πλευρά σας ώστε να μπορέσουμε να ε, διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα διότι είμαι βέβαιος ότι εν τέλει αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η γνωμοδότηση να τα ανακλά την πραγματικότητα και τα πραγματικά συμφέροντα των Ευρωπαίων Γεωργών και όχι να γίνει ε, απλώς ένα ε, προστατευτικό ε, κείμενο το οποίο δεν θα βοηθήσει κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όντως, είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση θα πρέπει η γνωμοδότηση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να αντανακλά την πραγματικότητα και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γεωργών. Περί αυτού πρόκειται θα πρέπει να διαφυλάξουμε κάποιες αξίες ε, και να δούμε τις τάξεις μεγέθους και τις διαφορές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα γίνει μια σειρά διμερών διαπραγματεύσεων που το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος κάποιο κλάδο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια το συνολικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους εκπροσώπους της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου που είχαν την καλοσύνη να έρθουν στη συνεδρίαση για να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Είναι σημαντικό όταν μιλούμε για το μοντέλο του, το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, να δούμε και τη, την κλίμακα, την τάξη μεγέθους, ε, τις ε, διαφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Αυστραλιανής Γεωργίας, Αυστραλέζικης Γεωργίας και αυτές τις διαφορές να τις λάβουμε υπόψη ώστε να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες. Ο κύριος Ταραμπέλα. Εγώ θα συνεχίσω από το συμπέρασμα του κυρίου Φιέλνερ και θέλω να πω σε όλους ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να συγχαίουμε την αναδίπλωση και τον προστατευτισμό. Προστατευτισμός μπορεί να είναι θετικό, ενώ η αναδίπλωση και το κλείσιμο στον εαυτό σου είναι κακό. Αλλά θα πρέπει να προστατεύουμε κάποιους βασικούς τομείς. Εάν προσθέσουμε όλες ε, τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν και γεωργικό σκέλος, είτε ε, ΣΕΤΑ με το Καναδά, είτε TTIP με τις ΗΠΑ, είτε και συμφωνία με το Μερκοσούρ, που εκεί ε, ο τομέας του βοηού κρέατος είναι πολύ ευαίσθητος, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, πέντε μεγάλους ε, ε, παραγωγούς παγκόσμιους ανέφερα σε προϊόντα γεωργικά. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, εμείς από όλους αυτούς τους μεγάλους ε, φορείς είμαστε εκείνοι που προστατεύουμε λιγότερο τους παραγωγούς μας σε όλους τους τομείς, γιατί απορριθμίζουμε τις αγορές, τώρα είμαστε έρμεα των παγκοσμίων τιμών. Εμείς απορριθμίζουμε τις αγορές μας, άρα υποβάλλουμε σε μια ξέφρενη όλο και περισσότερη μορφή ανταγωνισμού τους γεωργούς. Τι νόημα έχει να εισάγουμε κρέας από την Αυστραλία. θέλουμε να εφαρμόσουμε ε, τη Συμφωνία για το Κλίμα, θα πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε από το, την άκρη ε, του κόσμου ε, κρέας. Αυτό είναι ο προστατευτισμός και εγώ τολμώ να το ξεστομίσω, είμαι μόνος μου, αλλά δεν πειράζει, αναλαμβάνω τις ευθύνες. Έπρεπε να αρχίσω από εκεί, συγγνώμη, ε, να μιλήσω για τον εισηγητή. Ο Ρίκα Αντριώη, ε, τονίζει τα σημεία που είναι κίνδυνος για τη δική μας γεωργία. Ε, θα ήθελα να πω ότι ε, θα ζητήσουμε, να προσκαλέσουμε από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία μεγάλη διαπραγμάτευση να βάλει τη γεωργία ως πρώτο κεφάλαιο και όχι τελευταίο που πέφτει θύμα μετά στην προσαρμογή των άλλων πολιτικών. Και να πω και κάτι για τον Brexit τελειώνοντας. Το Brexit είναι πολύ περίπλοκο θέμα. Δεν γνωρίζω την κατάσταση στην Αυστραλία, καλύτερα γνωρίζω τα θέματα της Νέας Ζηλανδία. και όταν διαπραγματεύτηκε το 1973 την ένταξή του το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατάφερε να περάσει συγκριτικά πλεονεκτήματα και πρόσβαση στην αγορά των χωρών τη κοινοπολιτεία. Βλέπει Νέα Ζηλανδία για το πρόβιο. Ε, ρωτώ, εκείνα τα πλεονεκτήματα τότε που διαπραγματεύτηκε και επέτυχε το Ηνωμένο Βασίλειο ισχύουν ακόμα μετά το Brexit γιατί θα μας εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά ειλικρινή ερώτηση κάνω και θα παρακαλούσα και θα επιθυμούσα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο κύριο Ταραμπέλα έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί μερικές φορές στις διαπραγματεύσεις αναβάλλονται τα, γεωργα, γεωργικά θέματα και μετά βρισκόμαστε προ το τελεσμένο γεγονότων και μετά διαρριγνύουμε τα ημάτια μας και λέμε πώς συνέβη αυτό. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη γεωργία και να μην αναβάλουμε τα γεωργικά θέματα για το τέλος των διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το επισημάνουμε στον Επίτροπο γιατί πολλές φορές έχουν γίνει σημαντικές παραχωρήσεις προς εμπορικούς εταίρους εις βάρος της γεωργίας. Και πολύ εύστοχο το αποτέλεσμα του προλαλήσαντος. Θα πρέπει να αντανακλά η συμφωνία την πραγματικότητα και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γεωργών. Και αυτό είναι ένα είδο ιδιόρυθμου προστατευτισμού, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα. Ευχαριστώ κυρία Σένορα. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω μια κοινή παρέμβαση και για τα δύο θέματα, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα πλεονεκτήματα ε, τέτοιων διαπραγματεύσεων είναι πάντα μονομερή και ευνοούν μόνο τους μεγάλους εξαγωγείς και πάντα γίνονται εις βάρος των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων που ε, θα υποχρεωθούν να πληρώνουν, να πολλούν κάτω του κόστους παραγωγής. Πολύ φοβάμαι ότι οι μικρομεσαίοι παραγωγοί μας και οι γεωργοί μας δεν θα κερδίσουν τίποτα με τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Επίση, ε, και οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα βγουν κερδισμένε από τέτοιε συμφωνίε. Θα καταστραφούν θέσει εργασία και επιχειρήσεις, ε, κάτι που είναι ει βάρο ε, της υπαίθρου. Επίσης, οι συμφωνίες αυτές επηρεάζουν αρνητικά και είναι και για το κλίμα, για τις κλιματικές αλλαγές γιατί πολύ συχνά προβληματιζόμαστε για τις κλιματικές αλλαγές. Πολύ, πολλές ανησυχίες εκφράζουμε, αλλά σε τελική ανάλυση προωθούμε και υπογράφουμε συμφωνίες που αντίθετα θα αυξήσουν τα αέρια του θερμακηπίου. Και θα θέσουν σε κυκλοφορία στον πλανήτη εμπορεύματα που εισάγουμε από την άλλη άκρη του κόσμου, από την άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ θα μπορούσαμε να ευνοούμε τα πιο ε, σύντομα κυκλώματα. Επίσης έτσι αυξάνεται η κατασφατάληση των ενεργειακών μας ε, πηγών και της ενέργειάς μας. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να υπογράφουμε τέτοιου είδους δυσμενείς εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Mm. Ναι. Κυρίες και κύριοι, πολλά άκουσα σήμερα για ευκαιρίες που δημιουργούνται, λέει, από τη συμφωνία αυτή για τη Γεωργία. Κανένας δεν τις ανέφερε συγκεκριμένα. Αγαπητέ συνάδελφοι, αν θεωρείτε τώρα ότι θα πρέπει να στέλνουμε είναι από την Ευρώπη στην Αυστραλία, πλήσωμε. Μήπως και βόηο κρέας από την Ιρλανδία να εξάγουμε στην Αυστραλία. Μα Καμία ευκαιρία δεν έχει η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Είναι τελείως ανεδαφικά αυτά και καθόλου ρεαλιστικά. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για το ελεύθερο εμπόριο, αλλά όχι κάθε συμφωνία ξεχωριστά για να εξαιρούνται τομεί. Θα πρέπει να δούμε τη Μερκοσούρ, την Αυστραλία, την Ζηλανδία από κοινού όλες συμφωνίες και η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα είναι ο μέγας χαμένος αυτή την υπόθεση, διότι δεν έχουμε την παραμικρή ευκαιρία ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας με αυτές τις χώρες. Και όποιος ισχυρίζεται εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία ε, έχει τώρα ευκαιρίες, αυτό ε, είναι εξαπάτηση των Ευρωπαίων Γεωργών. Μα τι νόημα έχουν όλα αυτά. Να στέλνουμε στην άλλη άκρη της γης ε, στους αντίποδες προϊόντα που έχουν και εκείνοι τα ίδια. Εντάξει, καλό το εμπόριο, δεν λέω, αλλά δεν ευσταθεί καθόλου από την οικολογική σκοπιά αυτό. Καταστρέφουμε τον πλανήτη. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Αντριέ, θα μπορούσε να είναι και οξύτερος. Αλλά το συμπέρασμά του δεν το καταλαβαίνω ότι καλό το εμπόριο. Άμα τα λες όλα αυτά θα πρέπει να είσαι συνεπής και να λες όχι δεν έχει νόημα. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια λογική. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε μάθει τίποτα από τα λάθη της ΣΕΤΑ και της TTIP αλλά συνεχίζουμε χαροπά να διαπραγματευόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω καθόλου αυτά τα πράγματα. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να επιμείνω ότι η Επιτροπή μας έχει ελάχιστες δυνατότητες ε, σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Το λέω για άλλη μια φορά γιατί δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν κάτι ή να εγκρίνουν κάτι είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Σε καμία περίπτωση η Επιτροπή Γεωργίας. Εμείς ε, κάνουμε συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, συζητήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους αφορούν ε, συμφωνίες για τη Γεωργία και τελικά δεν έχουμε καμία δυνατότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα εκτός και αν είμαστε μέλη στην Επιτροπή Ιντα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ε, αποτελεί ε, ανισότητα για την Επιτροπή μας και το λέω για άλλη μια φορά γιατί ε, κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να δώσει μεγαλύτερη εξουσία σε αυτή την Επιτροπή για να μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις εμπορικές συμφωνίες όπου διακυβεύεται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να πούμε και εμείς κάτι και να το συμμερίζεται και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Όσον αφορά τη συμφωνία με την Αυστραλία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αξιολόγηση επιπτώσεων. Δεν ξέρω αν έγινε αξιολόγηση επιπτώσεων ε, στους συγκεκριμένους τομείς. Προφανώς η Αυστραλία έχει μεγάλες δυνατότητες ε, σε θέματα βόηου κρέατος ε, και πτηνών και όπως είπανε και η πρόβιο κρέας, συγγνώμη, θεωρούνται ευαίσθητοι τομείς μαζί με τη ζάχαρη και άλλα προϊόντα όσον αφορά τον Ίνο που ανέφερε ο συνάδελφος από την Επιτροπή Ίντα, εγώ νομίζω ότι δεν πουλάμε ούτε λίτρο κρασί από πλευρά Ευρώπη ε, στην Αυστραλία γιατί είναι αδύνατο. Το είπε και ο κύριο ε, Χάουσλινγκ, συμφωνεί, διαφωνεί, δεν έχει σημασία, αλλά είναι αδύνατο να πουλήσει κανεί ε, έστω ένα λίτρο κρασί στην Αυστραλία. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προστατεύει απόλυτα τον τομέα του ίνου τη Αυστραλία και είναι αδύνατο. Αυτοί έρχονται εδώ με χαμηλέ με χαμηλές τιμέ και ανταγωνίζονται στον ευρωπαϊκό τομέα. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάποια στρέβλωση υπάρχει κάποια ε, ανισότητα γιατί οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλότερες από τις τιμές του ευρωπαϊκού κρασιού. Ε, και φυσικά είναι πολύ χαμηλότερη και η ποιότητα, αλλά δεν έχουμε καμία δυνατότητα να παρέμβουμε σε αυτό. Θα ήθελα να ξέρω όμως αν υπάρχει εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν έγινε αξιολόγηση επιπτώσεων ε, και Εάν αποφασιστεί ότι θα ακολουθήσουμε, θα συνεχίσουμε τι εμπορικέ συμφωνίε, η κυρία Μάλστρομ ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία και θέλω να πω κάτι γιατί το ανέφεραν και ο συνάδελφος Ταραμπέλα και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Το θέμα του προστατευτισμού. Να προσέχουμε με αυτόν τον προστατευτισμό. Εγώ δεν θέλω προστατευτισμό διότι ο προστατευτισμός που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ε, από την ε, ε, κυβέρνηση Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείες σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε επιτραπέζιες ελιές στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις συνέπειες ε, της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητά η κυβέρνηση Τραμπ για να μην επιτρέπει εξαγωγές από την Ευρώπη ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βοήθειες, ενισχύσεις προς τους νέους γεωργούς, το greening κτλ. Εάν λοιπόν στις 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει ψήφισμα από το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν το σύστημα της κοινή γεωργικής πολιτικής. ΚΑΠ, ε, Νέοι Γεωργοί, Greening και το σύστημα των ενισχύσεων. Ε, όλα αυτά λοιπόν ε, επηρεάζουν όλους αυτούς τους τομείς, όλα αυτά βρίσκονται στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ και εγώ φυσικά δεν είμαι με αυτή την πολιτική και με αυτόν τον τρόπο. Ε, στην Ευρώπη για πολιτικά κριτήρια προστατεύουμε τους ευαίσθητους τομείς μας και πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει ε, να πωλείται βόλιο κρέα στην Αυστραλία και να το πουλούμε ε, στην εσωτερική αγορά. Ναι, αλλά ο προστατευτισμός ποτέ δεν θα ε, είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσω προς υπεράσπιση αυτών τον οποίο πρεσβεύω, γιατί δεν πιστεύω ότι βοηθά και δεν ευνοεί κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Σπανίως κάνω τόσα σχόλια, αλλά αυτή τη φορά είμαι υποχρεωμένος. Καταρχήν θα σας παρακαλούσα να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, γιατί δεν είναι κεκλεισμένο το θηρόν, οπότε μπορούμε να συμμετέχουμε εκεί για να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Επίσης, για τα θέματα αυτά θα πρέπει να μιλούμε και στις πολιτικές μας ομάδες, γιατί οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται στη διάσκεψη των Προέδρων. Οπότε, αν δεν ε, το λάβουν υπόψη, δεν πείσουμε τις πολιτικές ομάδες. Εδώ δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν. Εμείς ε, είμαστε ήδη πεπισμένοι, αλλά θα πρέπει να πείσουμε τις πολιτικές ομάδες για να μεταφέρουν αυτό το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων που λαμβάνει τις αποφάσεις για την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Και πολύ συχνά τέτοιου είδου θέματα περνάνε ως ε, κατ' αρμοδιότητα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Δεν θέλουμε να επιρρύπτουμε ευθύνε, αλλά θα πρέπει να παρέχουμε όλο το φάσμα των πληροφοριών, ώστε και σε εθνικό επίπεδο να μπορούν οι βουλευτές να το παρουσιάζουν και να μην ξυπνούν οι ευαισθησίες μας μόνο ενώπιση των εκλογών. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των γεωργών και να έρχονται οι, σε επαφή οργανώσεις των γεωργών με τους βουλευτές τους, ώστε να τους ευαισθητοποιούν και να τους παρουσιάζουν το εύρος των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ παρακολούθησα τη συζήτηση αυτή με ενδιαφέρον και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είμαι πολέμιος των εμπορικών συμφωνιών, ούτε είμαι υπέρμαχος του προστατευτισμού. Αλλά στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες χρειάζεται προσοχή να μην είναι όλα εις βάρος ε, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας αυτά που συμφωνούμε και η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία είναι χώρε γεωργικής παραγωγής. Βρήκα μερικά στοιχεία. Ακούστε για την παραγωγή γάλακτος. Από το 2010 μέχρι το 2016 αυξήθηκε στη Νέα Ζηλανδία κατά 24% γαλακτοπαραγωγή, στην Ευρώπη μόλις 12%. Έχω και στατιστικές. Από το 2008 μέχρι το 2016 η εξαγωγή βουτύρου από τη Νέα Ζηλανδία προς την Ευρώπη αυξήθηκε μόλις κατά 5% προς την Κίνα 500% κατανοητό γιατί η Κίνα είναι πιο κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Αυτό που με ενοχλεί είναι το μονοπόλιο ε, ε, μιας γαλακτοκομικής ε, παραγωγής 95% της παραγωγής επεξεργάζεται ένα γαλακτοκομείο στη Νέα Ζηλανδία, είναι μονοπόλιο. Στην Ευρώπη, 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν μόλις το 36% της γαλακτοπαραγωγής και σε ό,τι αφορά το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, κατά μέσο όρο 420 ε, αγελάδες έχουν ε, οι ε, αγελαδοτρόφοι στη Νέα Ζηλανδία και εδώ 36 αγελάδες και δεν χρειάζονται και στάβλους. Βόσκουν ελεύθερα τα ζώα το χρόνο στα λιβάδια στη Νέα Ζηλανδία. Και βέβαια δεν έχουν κρατικές ενισχύσεις Νέο Ζηλανδοί για λαδοτρόφια, αλλά δεν έχουν ούτε Κομισιόν, ούτε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τους πρίζουν. Αυτό που συμβαίνει πούμε, στην Ευρώπη συνέχεια. Θυμίζω και μόνο την απόφαση του Επιτρόπου ότι στο μέλλον ε, ε στα ψυχανθή δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ε, κτλ., έχουν εξαγριωθεί, έχουν βγει από τα ρούχα τους οι Γεωργοί, όλο το καλοκαίρι αυτό μου λέγανε. Άρα, ε, ε, όταν κάνουμε εμπορικέ συμφωνίες κύριε Φιέλνερ, και εγώ ξέρετε ήμουν μέλος 10 χρόνια στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, θα πρέπει να προσέξουμε να έχουμε περιορισμό και ποσοστώσει ε, με συγκεκριμένο αριθμό τόνων. Φυσικά δεν μπορούμε να περιχαρακωθούμε και να κλειστούμε στον εαυτό μας να τηρούνται όμως οι ποσοστώσεις Επίση, Ε, πρέπει να σας πω ότι ο συνεταιρισμός μου ήθελε κάποτε να πουλήσει τυρί στην Αυστραλία. Τράβηξε τα πάνδυνα και δεν θέλουν ούτε να το ξανακούσουν ούτε να το ξανακάνουν. Και ό,τι αφορά, ε, αφορά σε αυτά που είπε η συνάδελφος Αγγιλέρα, ο προστατευτισμός όχι μόνο δεν μας βοηθάει, αλλά ε, απειλεί και πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και κοιτάξτε, μια σύμπτωση περίεργη τώρα. Φαίνεται να συμφωνούν ε, διάφοροι ε, τύποι μεταξύ τους, όπως είναι η Greenpeace, άλλες ε, ΜΚΟ και ο πρόεδρος των ο κύριο Τραμπ. Ε, δεν θα πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες, να κάνουμε μια λογική συμφωνία με συγκεκριμένες ποσοστό. Ευχαριστώ. Κυρία Νόχλ. πάρα πολύ για αυτά που λέει ο κύριος Ντες, να μην έχουμε ελέγχους ε, και καθόλου κρατικές ενισχύσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Ε, πολύ ενδιαφέρον να τα πείτε και στους αγρότες αυτά. Ε, κοιτάξτε τι θέλω να πω. Ε, όταν συζητάμε ένα θέμα θα πρέπει να μιλάμε για την ουσία, για τα σημαντικά. Ποια είναι η ουσία. Έχει νόημα να ανταλλάσσουν δύο ήπειροι παρόμοια προϊόντα και δύο ήπειροι που δεν είναι μία δίπλα στην άλλη, αλλά είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν υπάρχει πιο μακριά από την Αυστραλία. Λοιπόν, έχει νόημα αυτό, πραγματικά αυτό αμφισβητώ, την ουσία την ίδια στο μέλλον και θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό. Δεν θα έχουμε ούτε το πετρέλαιο, ούτε τα καύσιμα για να κάνουμε αυτό το εμπόριο και κάποια στιγμή θα έχουμε φτάσει και στα ωριά μας. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω επί της ουσίας, για ποιο λόγο θα πρέπει να ταξιδεύει το βόηο κρέας από τη μία άκρη της γης στην άλλη και τούμπαλη. Και ακόμη για το τυρί. Και αρχίζουν ορισμένοι να χαίρονται και γυαλίζουν τα μάτια τους, θα εξάγουμε τυρί στην Αυστραλία. Ε, μα για να ε, φτιάξουμε τυρί θα πρέπει να φέρουμε σόγια από τη Βραζιλία, ε, όπου υλοτομούνται δάση για να σπαρεί η σόγια, ε, δάση που τα χρειαζόμαστε για την κλιματική αλλαγή, έρχεται εδώ για να εξάγουμε εμείς ε, τυρί στην Αυστραλία. Και τι θα μείνει η κοπριά στην Ευρώπη. Και το ευγενές προϊόν τυρί θα εξάγεται. Στη Γερμανία έχουμε πρόβλημα με τον υδροφόρο ορίζοντα. Η ΙΝΤΑ, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, τα συζητάει αυτά, τα σκέφτεται. Για ελάτε και σε κανένα αγρόκτημα να δείτε τα υπολείμματα και την κοπριά και δεν μιλώ για μια κανονική παραγωγή, μιλώ για υπερεντατική παραγωγή. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα που είναι και η ευημερία των ζώων με διάφορα πρότυπα και ε, υποχρεώσεις. Στο μέλλον θα τηρηθεί αυτό και την οικολογία και το κλίμα και την προστασία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εμένα με ενδιαφέρει κατά πόσο έχει νόημα. Δηλαδή, επειδή μπορώ να εξάγω στην Αυστραλία, θα το κάνω κιόλας, ε, έχει νόημα η δικιά μας γενιά δεν είναι ίδια με τη γενιά των γονέων μας. Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με διλήμματα, με πράγματα που είναι εφικτά, αλλά είναι και σκόπιμα, είναι και λογικά. Τώρα θα κάνουμε τέτοια ανταλλαγή προϊόντων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αποκρούσω την κατηγορία της κυρίας Νόιχελ που είπε ότι είμαι κατά των κρατικών ενισχύσεων για τους αγρότες. Πραγματικά για να μου προσάψει κανείς κάτι τέτοιο ε, χρειάζεται να είναι πάρα πολύ κακός. Έτσι και αλλιώς δεν τα παίρνω σοβαρά αυτά που λέει η κυρία Νόιχελ. Κύριε Χόιμπουχ, τώρα ποιος παίρνει ποιον στα σοβαρά, ας μην μπούμε σε τέτοια θέματα καλύτερα. Ας παραμείνουμε στην πραγματικότητα και στην ουσία. Έχει δίκιο η Μαρία Νόχελ. πές από το στόμα μου τα πήρε και με την καρδιά μου. Τι νόημα έχει για προϊόντα που παράγουμε οι ίδιοι και παντού στον κόσμο παράγονται αυτά τα προϊόντα. Μα είπε ο συνάδελφος από την Ίντα ότι έχουμε κακό εμπορικό συζύγιο για τον Ίνο, ας πούμε. Πόσο κρασί πια εξάγουμε από την Αυστραλία και ε, πόσο εισάγουμε ακόμα και αν καταργήσουμε όλα τα εμπόδια και να μπορεί να ρέει ο ίνος όπως θέλουμε. Στην Αυστραλία είναι κάπως λιγότεροι καταναλωτές. Ποτέ δεν θα έχουμε κελισμένο ισοσκελισμένο ισοζύγιο θα πρέπει να σκεφτούμε τι παράγουμε πού, για ποια αγορά και τι έχει νόημα να εμπορευόμαστε και να έχουμε και μια συνεκτική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Τα είπε πολύ ωραία η Μαρία Νόχελ και άλλοι συνάδελφοι. Για τις ποσοστώσεις τώρα και τους τόνους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι αν προσθέσουμε τις συμφωνίες με Αυστραλία και ε, Νότια Αμερική για το βόλιο κρέας συγκεκριμένα και ανοίξουμε και επελευθερώσουμε την αγορά μας, θα έρθουν επιπλέον 365.000 τόνοι. Μα τώρα έχουμε ξεχυλήσει από βόλιο κρέας. Θέλουμε ακόμα 365.000 τόνους στην Ευρώπη να εισάγεται. Ο συντάξης νομοδότης ο κύριος Αντριού έχει ε, γράψει μια πολύ καλή γνωμοδότηση, έχει εντοπίσει τα προβλήματα. Σε εμά τώρα εναπόκειται από κοινού να δράσουμε υπεύθυνα και πάντα να λέμε ποια είναι τα προβλήματα. Αλλά δεν έχει νόημα να απαριθμούμε όλα τα προβλήματα και τέλος να λέμε καλά δεν πειράζει, ας υπογράψουμε τώρα. Η γεωργία είναι πολύ σημαντική και για το κλίμα και για την ε, προστασία του και δεν νομίζω ότι υποφέρουμε από έλλειψη ποιοτικών τροφίμων, ούτε από επιλογή στην Ευρώπη. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε και θα ήταν πολύ μεγάλο το κέρδος και για τους καταναλωτές μας. Να σταματήσουμε αυτά τα πηγενέλα των εμπορευμάτων που, των τροφίμων που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μιλήσουμε στους καταναλωτές για την ποιότητα των τροφίμων, γιατί οι καταναλωτές δεν είναι πάντα ενήμεροι. Θυμάστε τι έγινε με το σάπιο κρέας, ε, τις αγωγές σάπιο κρέατος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και κοινοποίησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, της Ευρώπης και αλλού το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε και την επικοινωνιακή μας πολιτική και την σωστή ενημέρωση του καταναλωτή. Βέβαια, ε, το εμπόριο ε, είναι διμερές, δεν γίνεται πρώτα προς μια κατεύθυνση, δεν είναι σήμαντο. Ευχαριστώ, ο κύριος Δενανό. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και είναι αλήθεια ότι χωρίς να είναι κανείς κατά κατά των εμπορικών συμφωνιών, έχει παρόλα αυτά το καθήκον να προστατεύσει ε, τη, τη γεωργία και ιδιαίτερα στα πλέον, ε, στις πλέον ευαίσθητες περιοχές. για το πρόβλημα είναι η σώρευση όλων αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Έχουμε την συμφωνία Μερκοσούρ, ΣΕΤΑ και άλλες εμπορικές συμφωνίες. Ε, έχουμε στον ορίζοντα και την συμφωνία με το Βιετνάμ και άλλες χώρες. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα για τα πιο ευαίσθητα εδάφη. Μια στιγμούλα, μια στιγμούλα. Έκανα λάθος. Ήθελα να σα δώσω το λόγο στο τέλο μια και αντικαθιστάτε τον κύριο Αντρία. Ας ολοκληρώσουμε πρώτα τον κατάλογο των ομιλητών και μετά σε εσά, ο κύριος Φλάναγκαν. Thank you. I was just being The man wanted to talk. Εγώ απλώ ευγενικό είμαι, ήθελε να τα πει ο συνάδελφο. Αυτό το οποίο ε, προέχει στην Ολομέλεια για την κλιματική αλλαγή είναι ότι ε, κάθε φορά που περνάμε φαίνεται να γκρεμίζεται η ε, οροφή. Μετά πηγαίνουμε στις ε, επιτροπές μας και ακούμε τις διάφορες πιθανές εμπορικές συμφωνίες και ξεχνάμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει στην Ολομέλεια. Πώς γίνεται να τα κάνουμε και τα δύο. είναι ότι η αριστερά δεν ξέρει τι πει η δεξιά. Ε, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουν πει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και τελικά θα βάλουμε το βόλιο κρέας ε, στα σκάφη, θα διασχίζουν τον Ατλαντικό να συναντιούνται και τελικά όλα θα είναι καλά. καλώ καμωμένα. Ε, αυτά κάνουμε, βέβαια δεν αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα ένα από τα πράγματα ε, τα οποία υποτίθεται ότι θα προκύψουν είναι η αύξηση του ανταγωνισμού. Μου λένε ότι ο ανταγωνισμό οδηγεί σε καινοτομία και οδηγεί και σε βελτιώσει ε, τρόπων την δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε βελτιώσεις, ε, μηχανές παραγωγής γάλακτος, ρομποτικές κλπ. Αλλά τέλος πάντων, μπορούμε να παράγουμε μέχρι ενό σημείου ε, θα είναι όλο και πιο φθηνό, μετά θα ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να γίνεται φθηνότερο και τελικά ο παραγωγός δεν θα παίρνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε καινοτομήσει πάρα πολύ ε, με αυτόν τον τρόπο και η καινοτομία είναι πώς μπορούν να ζουν οι γεωργοί στην Αυστραλία και στην Ευρώπη με τίποτα και οι πολυεθνικές να κερδίζουν ε, τεράστια κέρδη. Ακούμε πάρα πολλά λόγια, όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή, τα συζητάμε μετά τη κλιματική αλλαγή και μετά κάνει τελείω διαφορετικό. Όλο λόγια ακούω και ανησυχία, ψευδή ανησυχία πρέπει να πω, για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Το συζητούμε στην Ιρλανδία, το συζητούμε εδώ και αρκετά χρόνια, το γνωρίζω γιατί ακούω το BBC συχνά ε, και τώρα το συζητούν πολύ και στη Μεγάλη Βρετανία. Και από ό,τι φαίνεται κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Και ένα από τα πράγματα που λέμε ότι θα κάνουμε είναι ότι θα συζητάμε τα προβλήματά μα τα συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε με τον γείτονα για να δούμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τα το ζήν γιατί ο ανταγωνισμός οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς στην αυτοκτονία. Αφού τα συζητήσουμε λοιπόν και καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και πάλι δεν μπορείς να επιβιώσεις και αυτή είναι η στρατηγική αυτή τη στιγμή για την ψυχική υγεία. Απλώς να τα συζητάμε. Ίσως θα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Μήπως ε, ε, θα έπρεπε να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να ανταγωνίζονται σαν τα σκυλιά, αλλά να είναι άνθρωποι που θέλουν ποιότητα ζωή, που θέλουν κάτι για ε, να πληρώνονται για αυτό που παράγεται. Και αυτό που θα κάνουμε εδώ ε, είναι να μην αυξήσουμε τα εισοδήματα των ανθρώπων, θα πάνε τα χρήματα στι πολυεθνικέ και θα έχουμε περισσότερα χρέη και περισσότερε αυτοκτονίε. Όπω είπε και μια ε, εθνική εφημερίδα, ο Independent, η Αυστραλία ουσιαστικά οδηγεί σε όλο και χαμηλότερε τιμέ γάλακτο και ένα άνθρωπο αυτοκτόνησε στην Αυστραλία γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει αυτά τα πράγματα. Ψηφίστε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θυμάστε τι θα προκαλήσετε. Θα προκαλήσετε άγχος, ε, στρες και θα κάνετε τους ανθρώπους μίζερους. Ε, εμείς δεν είμαστε πόροι, είμαστε άνθρωποι και πρέπει να μπορούμε να ζήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντερκάντελερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κανονικά, ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ παίρνει από τους πρώτους το λόγο σε τέτοιες συζητήσεις. Δεν πειράζει, καλά που αφήσατε τους άλλους γιατί παρακολουθήσαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πραγματικά διχασμένη η Επιτροπή μας και δίστανται απόψεις. Αν υπάρχει μια κοινή διαπίστωση, αυτή είναι η σημασία της γεωργίας σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Θα πρέπει να υποστηρίζετε και να υπογραμμίζετε. Το κείμενο του συναδέλφου Αντριού, όπως μας παρουσιάστηκε, ε, μας κάνει να πιστεύουμε ότι η Αυστριαλία εξάγει μόνο γεωργικά προϊόντα και καταλήγει προσοχή, προσοχή. Αυτό μπορεί να ισχύει μέχρι κάποιο σημείο, αλλά ε, πρέπει να το διορθώσουμε λίγο. Είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες εκεί η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Δεν είναι μόνο τα γεωργικά προϊόντα, 10% μόνο είναι τα γεωργικά προϊόντα που εξάγουμε. Υπάρχουν άλλα προϊόντα με θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Με ανάλυση κατά τομέα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, χρειάζεται διαφοροποίηση. Τα στοιχεία τα έχουμε όλοι, τα κοιτάξαμε. Αρέσουν στους αυσαλούς τα καλά μας προϊόντα. Ε, το, ε, τυρί, ελαιόλαδο, χοιρινό, κρέα, σοκολάτα και πάει λέγοντας. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, βεβαίως να λάβουμε υπόψη αυτά που είπε εκεί η κυρία Αγγιλέρα, να είμαστε επιθετικοί όπου χρειάζεται και αμυντικοί επίσης όπου χρειάζεται. Και θα επανέλθω στη συνέχεια για το κείμενο για τη Νέα Ισλανδία. Αν οι σκιώδεις είχαν ε, δηλώσει ότι θέλουν το λόγο στο πρώτο τμήμα, θα τον έπαιρναν και νωρίτερα. Αλλά αν το ζητούν ε, εκ των υστέρων, ε, δεν θεώρησα ότι πρέπει να τους δώσω το λόγο πριν τους άλλους συναδέλφους. Από την αρχή, αν δεν είχατε ζητήσει το λόγο, δεν το λαμβάνετε πρώτος. Ευχαριστώ, κυρία Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ. Ήδη πολλά είπαν οι συνάδελφοι και να σας επαναφέρω στο κυρίω θέμα της έκθεσης. Θα πρέπει να δώσουμε τη γεωρική προοπτική σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Δεν θα ψηφίσουμε υπέρ ή κατά τη συμφωνίας με την Αυστραλία. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό και κάνοντα την απλασίωση, θα πρέπει να δώσουμε την προειδοποίηση και την ανησυχία της Γεωργικής Επιτροπής, Επιτροπής Γεωργίας, όπως τη διατυπώνει ο εισηγητή, ο συντάκτη γνωμοδότησης και από τις συμπληρώνει συνάδελφοι. Υπάρχουν ε, προβλήματα στην παράγραφο 3 και 4 για τα ευαίσθητα προϊόντα. Αυτέ οι ανησυχίε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά υπάρχουν και ευκαιρίε και ο κύριο Φιέλνερ τόνισε αυτό το τη συζήτηση. Οι Ευκαιρίε που δημιουργούνται με τη Νέα Συμφωνία. Το θέμα του περιβάλλοντο, των κλιματικών αλλαγών και πρόσβαση στο νερό. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα θέματα αφορούν την παγκόσμια γεωργία, όχι μόνο την ευρωπαϊκή είναι παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργία παγκοσμίω και θα επηρεάσουν και τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Ό,τι αφορά την παράγραφο 7, ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν κατάλαβα καλά σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις εμπορικές συμφωνίες ή την πιθανή συζήτησή του στο μέλλον, γίνεται σε επίπεδο 28 χωρών μελών, γιατί το Brexit δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οπότε προβληματιζόμαστε και ανησυχούμε τι θα γίνει μετά τη διεκπαιρέωση του Brexit, τι θα γίνει με τις συμφωνίες αυτές. Δεν ξέρω αν μπορεί από τώρα να το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως σκόπιμο θα ήταν να το κάνει κάποια στιγμή. Πάντως από άποψη γεωργίας εκφράσαμε κάποιες ανησυχίες για τη συμφωνία με το Μερκοσούρ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού στις συμφωνίες αυτέ. Εγώ δεν είμαι κατά των εμπορικών συμφωνιών εξορισμού. Πάντω θεωρώ ότι ω Επιτροπή Γεωργίας έχουμε καθήκον να γύρουμε τι ανησυχίε μα για τα ευαίσθητα προϊόντα, ώστε όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσει τη διαπραγματεύση να έχει υπόψη τι αυτέ τι ανησυχίε και να τι λάβει υπόψη με τρόπο που δεν θα παρεμποδίζουν, θα παραβλάπτουν, ε, θα, θα ζημιώνουν τη γεωργία στην Ευρώπη που διέπεται από την κοινή γεωργική πολιτική που επίση υφίσταται πιέσει. Ελπίζω λοιπόν να δώσει απαντήσει στις απορίε που έγινε η έκθεση και θα καταθέσω και εγώ κάποιε τροπολογίε στη γνωμοδότηση του κ. Αντρία. Ε, εγώ έγινα μάρτυρας αυτή τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και ε, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική καλύπτει ε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι διμερείς τριμερείς συμφωνίες ε, παρόλα αυτά επηρεάζουν ε, ε, την παγκόσμια γεωργία. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση. Και εκεί έγκυται και η δυσκολία των διαπραγματεύσεων μερικές φορές. Ο κύριος Άγνιου. Σας ευχαριστώ. Χθε μου τηλεφώνησα κάποιο από την πρεσβεία τη Αυστραλία, δεν είχα το χρόνο να το μιλήσω εκτενώς, αλλά μου έστειλε ένα ενημερωτικό σημείωμα και τώρα γίνονται δύο συζητήσει παράλληλα. Η μία αφορά την εμπορική συμφωνία με την Αυστραλία και άλλη με τη Νέα Ζηλανδία. Και φαντάζομαι όσοι λαμβάνουν το λόγο θα τον ξαναζητήσουν αργότερα. Το ίδιο ισχύει για μένα. Οι Αυστραλέζοι έχουν πρόβλημα με το ύφο των αρχικών παραγράφων, γιατί για τη Νέα Ζηλανδία μιλούμε για φιλόδοξη, ισορροπημένη και περιεκτική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Για την Αυστραλία όμως είναι διαφορετικό το ύφος και η διατύπωση. Λέμε ότι έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό τομέα με εξαγωγικό προσανατολισμό στην Αυστραλία. Εδώ δίνεται έμφαση στην αμυντική πτυχή. Ε, πάντως, ε, ένας από τους δύο μιλητές στην πρωινή συζήτηση μας εξήγησαν ε, γιατί θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, και γιατί δεν είναι εύκολο να ε, πουλήσουμε ευρωπαϊκό ίνο στην Αυστραλία και δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, όσο φαίνεται. Ε, και αφορά το θέμα των μη δασμολογικών φραγμών και τέτοιο θεμάτων. Πάντως, εγώ θα ξαναμιλήσω με κάποιον από την Αυστραλινή Πρεσβεία και θα του ε, θα το ρωτήσω λεπτομεριακά για όλα αυτά τα θέματα και σας προσκαλώ όποιον ενδιαφέρεται να έρθει στο γραφείο μου να το κάνουμε από κοινού. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάκριση βάρους Αυστραλίας και όχι της Νέας Ζηλανδίας. Και με τις εμπορικές συμφωνίες με τις δύο χώρες θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τον αντίκτυπο του Brexit που επίση είναι σημαντικός. Γιατί ε, ακριβώς ένα τρίτο των ε, εξαγωγών της Νέας Ζηλανδίας πηγαίνει προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Εξού και έλλειψη ισορροπίας και η έλλειψη δοσμολογικών ποσοστώσεων. Και επίση δεν εξαντλούνται όλε αυτέ οι δασμολογικέ προστώσει, γιατί έχουν αυξηθεί οι εξαγωγέ προ την Ανατολική Ασία, μια τεράστια αγορά και μάλιστα πολύ πιο κοντά. Οπότε νομίζω ότι ο πραγματικό φόβο, η πραγματική κατάσταση είναι πολύ λιγότερο ανησυχητική από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση. Γιατί η νοτιοανατολική αγορά επεκτείνεται με ταχύτητα του ρυθμού και φυσικά είναι πολύ, εύκολη, πολύ πιο εύκολη πρόσβαση των δύο χωρών, Νέα δηλαδή και σε αυτή. Επίσης, η Νοζηλανδία και η Αυστραλία Γεωργία δεν είναι τεράστιοι γεωργικοί όμιλοι, είναι περισσότερο οικογενειακέ και μικρέ εκμεταλλεύσει. Και υπάρχουν γεωργοί που δραστηριοποιούνται χωρίς καμία κρατική ενίσχυση. Πάντως οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξημένο κόστος λόγω και της υπερβολικής νομοθεσίας. Η ID για παράδειγμα, αυτή το, το σύστημα μεμονωμένης και ηλεκτρονικής ταυτότητας των προβάτων θα είναι υποχρέωση των κτηνοτρόφων να το κάνουν και είναι δαπανηρή διαδικασία. Οι Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί κτηνοτρόφοι δεν υποχρεούνται σε τέτοιο σύστημα και μπορούν να πολλούν το, το, το, κρέα του εδώ. Επίση, έχουμε ε, ζώνε απαλλαγμένε από νητρορύπανση. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Οπότε η ικανότητά μα να διαχειριζόμαστε τη γεωργία όπω θα θέλαμε περιορίζεται από τα κοινοτικά μέτρα. Επίση έχουμε και ε, την απαγόρευση πια να θάβουμε το, τα θανατωμένα μας ζώα στην, ε, κοντά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Τώρα έχουμε υποχρέωση να τα αποτεφρώνουμε. Ε, φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να θάβουμε από το να αποτεφρώνουμε τα ζώα, θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Επίσης, με τα δόντια των ζώων και πότε κάποιες υποχρεώσεις που ισχύουν ε, για, τη, για την ε, προβατοτροφία στην Ευρώπη που δεν ισχύουν αντίστοιχα στην ε, Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οπότε, αν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά και, και να πηγαίνετε σε σούπερ μάρκετ και να αγοράσετε μόνο ευρωπαϊκά προϊόντα και να δακτυλοδεικνύετε όσους δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η τακτική θα πρέπει να ακολουθήσετε αν θέλετε να είστε συνεπείς. Η χνηλασιμότητα είναι ε, πολύ σημαντικό θέμα και τη διεκδικούν και οι καταναλωτές και είναι σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και για τα προϊόντα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Σας ευχαριστώ. Όπως διαπιστώσατε δεν σας περιορίζω στο χρόνο αγόρευση αλλά θα ήθελα να επιδείξετε εσείς ήδη μια αυτοσυγκράτηση. Ο κύριος Βαλκάρ Σελσίσο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν ε, θα επισέλθω τώρα σε συζητήσεις. Ε, ορισμένες φορές ε, η αντιπαράθεση φαίνεται να είναι υψηλότερη της λογικής και δεν, δούμε, δεν βλέπουμε το συλλογικό συμφέρον των γεωργών, που είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η γεωργία δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς αντάλλαγμα ισοτιμία για τις εμπορικές συμφωνίες. Γιατί θα πρέπει ε, πριν από κάποια πρόταση να αναλύσουμε όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές τις συμφωνίες ε, σε τομείς όπως είναι το κρέας, ε, τα δημητριακά ή τα γαλακτοκομικά, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο εισηγητής στο σημείο 4. Φαίνεται επίσης ότι είναι άκρος απαραίτητο να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ε, γεωργούς τα αμύγδαλα, διότι εκεί πρέπει να γίνει διάκριση με τα προϊόντα ε, ε που προέρχονται από εκεί, διότι σε θέματα ποιότητας τουλάχιστον πρέπει να γίνεται η διάκριση σε αμύγδαλα, σε σπεριδοειδή, σε ίνο, σε τέτοια προϊόντα. Πάντα εμείς έχουμε προϊόντα αριστείας σε ευαίσθητου λοιπόν τομεί και στις γεωγραφικές ενδείξει, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει πριν υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία. Και ε, πέραν αυτού θα πρέπει να ακολουθήσουμε ανοιχτή γραμμή ε, στις αγορές που είναι η γραμμή την οποία εντείναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε ανταγωνιστικά προϊόντα όπως για παράδειγμα τα φρούτα με ε, καρπό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν την ευαίσθητη συμφωνία, την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν λόγω του εμπάργου με τη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να προωθούμε μέτρα, όπως για παράδειγμα απόσυρση κάποιων προϊόντων και εκστρατείες προώθησης κάποιων προϊόντων. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, έκανα μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή ημέρα φρούτων, που την υποστήριξαν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να υποβάλουμε ε, τροπολογίες για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε τουλάχιστον το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εμπορικές συμφωνίες ε, είναι σημαντικές ε, γιατί ανοίγουν νέες αγορές στα γεωργικά μας προϊόντα ε, και όταν έχουν προστιθέμενη αξία έχουν και νόημα. Όταν όμως αγκυμονούν κάποιους κινδύνους για τομείς που ήδη είναι ευαίσθητοι, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που εξέφρασαν ανησυχίες, αλλά διαπίστωσαν επίσης ότι ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, εμπορικές συμφωνίες συνάπτονται και δεν λαμβάνονται διόντως υπόψη παρατηρήσεις της Επιτροπής Γεωργίας θα έπρεπε σε τέτοιου είδου εμπορική συμφωνία ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι πιο ισχυρό. Γιατί εμεί ε, ε, έχουμε εκλεγεί άμεσα από του Ευρωπαίου πολίτε, ε, του εκπροσωπούμε και μεταφέρουμε τη δική του φωνή και τη δική του άποψη. Προσοχή λοιπόν και για τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη. Μέχρι στιγμή ούτε σε μία συμφωνία που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλε χώρε ή σε καμία διαπραγμάτευση που έχει γίνει, γιατί πολλές διαπραγματεύσεις έχουν ε, ξεκινήσει. Δεν έχουν περιλάβει ούτε μία, ε, ένα ε, κροατικό προϊόν με γεωγραφική ένδειξη, με ονομασία προέλευσης μάλλον. Ούτε σε μία εμπορική συμφωνία, ούτε σε μία εμπορική διαπραγμάτευση δεν έχουμε ούτε ένα κρατιόν με ονομασία προέλευση. Γιατί λοιπόν γίνεται κάτι τέτοιο, με ποιον τρόπο γίνονται οι επιλογέ. Γιατί και η Κροατία είναι εδώ και τέσσερα χρόνια ε, ε, 14 χρόνια μέλος, Ευρω... 4 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγιναν πολλές ε, συζητήσεις και συμμετείχαμε σε συζητήσεις για τις γεωρικές ε, διαπραγματεύσεις αλλά παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να συμπεριλάβουμε ούτε ένα προϊόν ε, κροατικό με ονομασία προέλευση σε τέτοιους συμφωνίες. Αυτό είναι διάκριση, διάκριση βάρους Κροατίας. Ο κύριος... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φιέλνερ για τη συνέπεια της σκέψης του γνωρίζουμε ότι ε, είναι αποφασισμένος να ανοίξει διάπλατα την ε, ευρωπαϊκή αγορά για να ε, εποφεληθεί όλων των προϊόντων που παράγονται ανά τον κόσμο. Αλλά αγαπητέ συνάδελφοι, η γεωργική παραγωγή δεν είναι βιομηχανική παραγωγή. Άλλοι μεταφέρεται, μετεγκαθίσταται, άλλοι υποκαθίσταται και άλλοι όχι. Άρα, ε, αν καταργήσουμε κάπου μια παραγωγή που είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, δεν έχουμε υποκατάστατο ή κάτι να την αντικαταστήσουμε. Υπάρχουν κάποια μέρη που έχουν συγκεκριμένη ε, βλάστηση, χορτολιβαδικές εκτάσεις και προσφέρονται μόνο για προβατοτροφία ή για βοοτροφία και αν εκεί ε, πνεύσουν ανεξέλεγκτα οι άνεμοι της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης θα ρημάξει ο τόπος. Θα εξαφανιστεί. Δεν επιτρέπεται αυτό να το κάνουμε. Μη τι άλλο για μια στοιχειώδη βιοπικιλότητα. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία είναι πλούσιες χώρες, είναι σπουδαίες χώρες από τις πλουσιότερες στον κόσμο και βεβαίω είναι ενδιαφέρον να έχουμε εμπορικέ συμφωνίε για κάποια βιομηχανικά προϊόντα και τι υπηρεσίε μα. Αλλά για τη γεωργία οι συνθήκε ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμού δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη. Λόγω τη δομή των γεωργικών μα εκμεταλλεύσεων. Λόγω και της μορφολογίας τη υπήρου μα, του εδάφους, ε, το κλίμα ε, ε, διαφέρει. Καμία σχέση δεν έχει με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Οι δύο αυτές χώρες ανέκαθεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και τη στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία ε, προετοιμάζεται να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μένα τουλάχιστον τυχοδιοκτικό να κάνουμε συμφωνίες με αυτές τις δύο χώρες. Αύριο η Μεγάλη Βρετανία κινδυνεύει να υπογράψει συμφωνία με τις παλιές τις κτήσεις που παραμένουν σήμερα στην κοινοπολιτεία και εμείς Ευρωπαίοι θα χάσουμε μια πολύ σημαντική αγορά. Θυμίζω τα στοιχεία για το κρέας. Η Μεγάλη Βρετανία εισάγει περίπου 2 εκατομμύρια τόνους κρέας, 700 εκατομμύρια τόνους μόνο από την Ιρλανδία. Και ε, μιλάω από τον έλεγχο της συναδέλφου Μαγκίνες. Αν μεθαύριο αποφασίσει η ε, Βρετανία ε, να τα βρει με Αυστραλία και Ζηλανδία που είναι χώρες κοινοπολιτείε, τι θα τους κάνουμε εμεί τους 2 εκατομμύρια τόνους βοηού που εξάγουμε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Και η διαπραγμάτευση αυτή, όπως και η διαπραγμάτευση με το Μερκοσούρ, για τα γεωργικά θέματα τουλάχιστον, δεν θα πρέπει να διακοπεί, αλλά να ε, μπει λίγο στην άκρη μέχρι να δούμε πού το πάει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το τι θα γίνει μετά την έξοδο. Εάν συνάψει εμπορικέ συμφωνίες, αν διατηρήσει τις ευρωπαϊκές μπορεί να έχουμε κάποια συμφωνία με Μερκοσούρ, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Εάν όχι, θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Δεν θέλω να κλείσω καμία πόρτα, αλλά μιλώ για την αρχή της προφύλαξης που θέλω να εφαρμοστεί για να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τη γεωργία ανεξαρτήτως παραγωγής. Γιατί το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τα τυριά, ε, για τα κρασιά, ωραία. Αν και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι στην Αυστραλία πολύ συχνά Ευρωπαίοι παραγωγοί και ε, συγκεκριμένα Γάλλοι έχουν πάει εκεί για να αναπτύξουν ε, τα μπέλια και τα κρασιά, να ε, φτιάξουν κρασιά παρόμοια με τα δικά μας για να είναι ανταγωνιστική ιδιαίτερα στην κινέζικη αγορά. Η κυρία Ντελαέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Θα ήθελα μόνο να επιμείνω εγώ στο γεγονός ότι Ευτυχώ που μπορεί να συμμετέχει στι συζητήσει για τις διμερεί συμφωνίε η Επιτροπή Γεωργία και καλά κάνουν και μας ρωτάνε. Θα πρέπει εμεί να έχουμε μια πάρα πολύ στεναρή θέση, ε, ε, θέση Ξέρουμε ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχει ανέκαθεν πιο φιλελεύθερες ε, τάσεις και στάσεις και θα πρέπει εμείς να συνεργαστούμε για να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία με την Αυστραλία. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Αντριέου για το έργο του. Οι προτάσεις του πραγματικά βαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ με το σύνολο των προτάσεων και το πάω ακόμα παραπέρα. Σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι το βόλιο και το πρόβιο κρέας, εγώ θα ζητήσω να εξαιρεθούν τελείως από τη διαπραγμάτευση. Γιατί από τη γεωργική σκοπιά Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία των ε, γεωγραφικών ενδείξεων, όπως ε, έγινε και με τη συμφωνία για τον Καναδά. Και τώρα... Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κλάρκ, ε, που ήταν από την αρχή παρόν. Ο διευθυντής ο κύριος Κλάρκ και μετά ο εισηγητής. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για αυτές τις δύο συμφωνίες, επομένως ε, σαφώς ευπρόσδεκτη η γνωμοδότηση και φυσικά συμφωνούμε ε, με την πλειοψηφία των όσων περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση του κυρίου Αντρία. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο εάν η γνωμοδότηση αναγνώριζε ότι υπάρχουν και κάποιοι ωφέλη για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη συμφωνία με την Αυστραλία. Δεν είναι μονομερή στη συμφωνία. Αυτό αναγνωρίστηκε, για παράδειγμα, στην περίπτωση του σχεδίου έκθεση για τη Νέα Ζηλανδία. Και ισχύει ακόμα περισσότερο για την Αυστραλία, που είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά από τον Καναδά. Ε, συμφωνώ ε, βεβαίως ε, με όσους ψήνουν ε, την προσοχή για ευαίσθητα προϊόντα στον γεωργικό τομέα στη συμφωνία αυτή, με την, διαπραγμάτευση μάλλον με την Αυστραλία. Και σίγουρα συμφωνούμε με τον κύριο Αντριέ και το βασικό μήνυμα που θέλει να διαβιβάσει, που ε, εξέφρασε και, σαν και πολύ εδώ, για τους πιο λεπτούς τομείς, ε, το βόιο κρέας, το πρόβιο κρέας, ε, αλλά επίσης τη ζάχαρη, το ρύζι. Σε όλους αυτούς τους τομείς η Αυστραλία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Όπως επίσης και ε, έγινε και με τη γνωμοδότηση με τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ε, περιχαρακώσουμε ευαίσθητους τομείς. Ε, δεν γίνεται μόνο μέσω απελοκλεισμού, αλλά και μέσω ποσοστώσεων στους δασμούς, μέσω μεταβατικών περιόδων, μέσω συγκεκριμένων δικλείδων ασφαλείας. Και επομένως δεν νομίζω ότι θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι θα έχουμε πλήρη αποκλεισμό στην Σύμφωνη Ελευθέρω με την Αυστραλία νομίζω ότι ε, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στη γνωμοδότηση στο συμπέρασμα, όπω γίνεται και με τη γνωμοδότηση για τη Νέα Ζηλανδία, ότι υπάρχει μια εργαλειοθήκη για να αντιμετωπίσουμε όλου αυτού του πιο λεπτού τομεί. Επίση, ε, συμφωνούμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο τη γνωμοδότηση που λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τι σορευτικέ συνέπειε ε, των εκχωρήσεων που γίνονται στι διάφορε συμφωνίε και να μην εξετάζουμε την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία μεμονωμένα. Σίγουρα θα το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι και η εντολή του Συμβουλίου το φθινόπωρο θα αντανακλά και αυτή ακριβώς ε, το ίδιο σημείο. Ε, κάποιες ακόμα παρατηρήσεις ε, για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που έθεσαν ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου. Στην παράγραφο 7 της γνωμοδότησης για το Brexit. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει οριστικοποιήσει την άποψή της ακόμα για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, το θέμα των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που θα ε, τεθούν σε ισχύ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το γενικότερο σκεπτικό ε, συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τη γνωμοδότηση του κ. Αντριέ. Δηλαδή ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη με τον ένα με τον άλλο τρόπο το γεγονό ότι μετά από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου η αγορά των 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιου τομεί, το βόλιο κρέα, το πρόβιο κρέα, για τη ζάχαρη θα είναι μικρότερη. Τέλος. Αρκετοί οι ομιλητές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής, ε, το περιβάλλον, ε, το υψηλότερο κόστος παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο αν η Επιτροπή Γεωργίας ε, στα πλαίσια αυτής της γνωμοδότησης, επισημάνει ότι αυτή η συμφωνία, όπως γίνεται και με όλες τις συμφωνίες, θα πρέπει να προσφέρει κίνητρα για βιώσιμη γεωργική ε, ε, παραγωγή, περιβαλλοντική βιώσιμη παραγωγή, υψηλέ ε, προδιαγραφές για την προστασία των ζώων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να πιέσουμε και τους εταίρους μας να καταλήξουν σε πολύ υψηλά πρότυπα και αυτοί. Αυτά λοιπόν ως απάντηση σε κάποιες από τις ανησυχίες και ιδέες που εκφράστηκαν στην αίθουσα θα μπορούσε αυτό ίσως να ε, αναφέρεται και στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, θα έχουμε φαντάζομαι ερωτήσει και στο δεύτερο τμήμα τη συζήτηση για την άλλη εμπορική συμφωνία, οπότε μπορεί να επανέλθετε και κύριε Διευθυντά. Ο κύριο Δενανό. Ευχαριστώ. Όντω, η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και έμεινα ικανοποιημένο με τη συμφωνία που εξέφρασαν οι περισσότεροι συνάδελφοι με τη γνωμοδότηση του κυρίου Αντριέ. Χωρίς ε, να είμαστε πολέμοι των εμπορικών ε, συμφωνιών. Έχουμε, πιστεύω, το καθήκον να προστατεύουμε τα εδάφη μας και τη γεωργική μας παραγωγή, ιδιαίτερα για τους ευαίσθητους τομείς. Γιατί, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, το πρόβλημα που τίθεται είναι η ισόρευση, ε, το άθροισμα όλων αυτών των ε, συμφωνιών. Μερκοσούρ, ΣΕΤΑ, θα έχουμε σύντομα Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ή με την Υποσαχάριο Αφρική. Επίσης, Διαπραγματεύσει με χώρες Μέσης Ανατολής. Οπότε αυτό άθροισμα όλων των εμπορικών συμφωνιών θα δημιουργήσει δυσκολίες. Επίσης, είχαμε ζητήσει έντονα μελέτη επιπτώσεων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να μας παρουσιάσει μελέτη επιπτώσεων για τις πιο ευαίσθητες γεωργικές παραγωγές. Ε, κυρίως βόηο και πρόβιο κρέας, αλλά και για το γάλα που ήδη βρίσκεται σε δίνη κατάσταση στην Ευρώπη. Και θέλουμε αξιόπιστα στοιχεία για να κάνουμε τις συγκρίσεις. Και θα πρέπει να έχουμε ε, μελέτη όχι μόνο για τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά και τον εδαφικό αντίκτυπο. Θέλουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες και ε, μελέτη του αντικτύπου όλων αυτών των ε, εμπορικών συμφωνιών και κυρίως του αθρίσματος, του σωρευτικού αποτελέσματος όλων αυτών των συμφωνιών στη γεωργία και τους άλλους κλάδους. Γιατί δεν μπορούμε επίση να έχουμε εμπορικέ συμφωνίε χωρίς να βρίσκεται η Γεωργία στην καρδιά των συζητήσεων και των ανησυχιών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Ήταν πραγματικά απλούσια η συζήτηση, χωρίς χρονικό περιορισμό στις αγορεύσεις. Μπορούμε τώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο ένα παρόμοιο με το προηγούμενο, γιατί αφορά τη σύσταση για τη διαπραγματευτική εντολή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νέα Ζηλανδία. Η συγητής μας, ο συντάκτης της γνωμοδότης είναι ο κύριος Νίκολσον. Και να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στην την 1η Σεπτεμβρίου στις 11 ώστε να εγκρίνουμε το σχέδιο γνωμαδότης 25 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα ψηφίσει στις 11 Οκτωβρίου και ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί πότε θα πάει η έκθεση στην Ολομέλεια. Περνάμε λοιπόν στη συζήτηση της έκθεσης του κυρίου Νίκολσον, της γνωμοδότης Νίκολσον, με παρεμφερές θέμα με το προηγούμενο, την εμπορική συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Περιμένουμε με ανυπομονησία λοιπόν την παρουσίαση του κ. Νίκολσον και φυσικά και τις τροπολογίες αργότερα. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των δύο συμφωνιών. Θα ακούσουμε λοιπόν τον συντάκτη της γνωμοδότης, τον κύριο Νίκολσον, για τη Νέα Ζηλανδία τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήταν σωστό και δίκαιο να πούμε ότι η συζήτηση αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την παρουσία του κυρίου Φιέλνερ, ο οποίος βέβαια στο μεταξύ έχει φύγει, για να ακούσει την Επιτροπή Γεωργία και τη γνώμη τη. Μπορεί να μην γνωρίζουν οι συνάδελφοι ε, το γεγονός ότι και ο κύριο Ανδριό και εγώ είχαμε λιγότερο από μία εβδομάδα για να ε, συντάξουμε τις νομοδοτήσει μας. Περίεργο, δεν είναι. Και λυπάμαι που έφυγε ο κύριος Φιέλνερ. Θα πρέπει νωρίτερα εμείς να έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε τις προτάσεις μας στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και στον κύριο Φιέλνε. Γιατί είναι αντίστοιχα τα προβλήματα και τα θέματα και δεν θα πρέπει να μας παραγωνίζουν και να μας λέει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ότι δεν έχετε κανένα λόγο, εσείς η Γεωργία είναι δική μας δουλειά και εσείς να μην ανακατεύεστε. Είναι και θέμα έτσι, πολιτισμού κοινοβουλευτικού. Ξέρω ότι ο κύριος ε, Κλάρκ δεν απάντησε στην ερώτησή μου την περασμένη φορά. Έχει μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες ως προς τα ποσά Δηλαδή πόσες ακόμα εμπορικές συμφωνίες θα κάνουμε μέχρι να βρεθούμε σε δινή θέση. Ακούσαμε ότι ε, αναφέρθηκε το πρωί συμφωνία Mercosur, είδαμε τι αντιμετωπίσαμε με το TTIP και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα εστιάζει συμφωνίες με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία γιατί η TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε απέθανε από την εκλογή του Donald Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε επικεντρώσει τώρα τις δυνάμεις, τις την ενέργειά μας και το προσωπικό μας σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και αλλού. Ε, πόσες εμπορικές συμφωνίες αντέχουμε ακόμα δηλαδή ε, μέχρι να κορεστεί η ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό ε, το έχω ξαναρωτήσει και το ξαναθέτω σήμερα. Ε, η Νέα Ζηλανδία είναι σε καλύτερη μοίρα από την Αυστραλία που έφαγε ξύλο σήμερα το πρωί γιατί ήταν πρώτη στην ημερήσια διάταξη. Μάλλον θα τη γλιτώσει η Νέα Ζηλανδία. Αλλά φαίνεται ε, ότι εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τις δύο αυτές χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναμένει να αρχίσουν σε λίγους μήνες και επίσημα οι διαπραγματεύσεις, φαντάζομαι μέχρι τα τέλη του έτους. Και είναι σημαντικό να πει τη γνώμη της και η Επιτροπή Γεωργίας. Δεν είμαστε κατά το, το ελευθέρω εμπόριο. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το είπε και ο κύριος Νταντάν προηγουμένως και η κυρία Αγγιλέρα. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση στην Επιτροπή Γεωργίας ότι δεν μπορούμε να ε, ζούμε σε ένα γυάλινο πύργο. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και είμαστε. Ε, αλλά μας θεωρούν ε, εμάς την Επιτροπή Γεωργίας προστατευτιστές. Όντως μας θεωρούν κάποιοι. Και θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ως προς την εικόνα που δίνουμε ε, προς τα έξω και τι μηνύματα στέλνουμε στο μέλλον. Πολλά από τα προϊόντα για τα οποία συζητούμε είναι εποχιακά. Και με ενδιαφέρον άκουσα όπως και ο κύριος Άγνιο ε, εξαγωγές ευρωπαϊκού ίνου. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ε, ένα θέμα προς διαπραγμάτευση. Λέτε ότι αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια οι εξαγωγείς. Μα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στις διαπραγματεύσεις αυτό. Η Νέα Ζηλανδία έχει πολύ διαφορετικό μοντέλο παραγωγή γεωργικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ ανταγωνιστική, ισχυρά εξαγωγική και είναι μικρή η γεωργική ενίσχυση είναι πολύ εκτεθειμένη στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ασταθείς και θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια μελέτη για τον πιθανό αντίκτυπο. Συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι ενδεχόμενες ε, ζημίες, απώλειες και τα κέρδη για τους ευρωπαίους παραγωγούς και τελικά ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε κάποιες παραχωρήσεις που κάνουμε στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να εξεταστούν πλήρως το πλαίσιο της πρόσβασης στην αγορά. Και θα πρέπει να εξεταστούν πλήρω λοιπόν στο πλαίσιο τη πρόσβαση στην αγορά που έχει ήδη χορηγηθεί βάσει του ΠΟΕ και άλλων εξελίξει διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το κάνει αυτό με επικοδομητικό τρόπο και είμαι βέβαιος ότι το κάνει με τους βασικούς ε, γεωργικούς φορείς να τηρούνται ενήμεροι για κάθε εξέλιξη σε σχέση με τη γεωργία. Μπορούμε να έχουμε μια δίκαιη και ε, καλή συμφωνία. Θα πρέπει ο ε, αγροδιατροφικός τομέας να θεωρείται εταίρος και όχι εμπόδιο στη συμφωνία μια φιλόδοξη συνολική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να προστατεύει τους ευαίσθητους τομείς Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, μπορεί να είναι προς όφελος και των δύο χωρών και να είναι ευκαιρία για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως ηγετική δύναμη στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρθιν ο πρώτος αυτό το γύρο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα θέματα που με απογοήτευσαν περισσότερο από τότε που έγινα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτό το οποίο θεωρώ αποτυχία αυτής της Επιτροπής πολύ συχνά να μπορέσει επαρκώς να σταθεί στο ύψος της και να δώσει μάχη υπέρ των αγροτών στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Και αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον και το είδα και όταν συζητούσαμε τη ΣΥΤΑ και το Μερκοσούρ και την DTIP στο παρελθόν, πολύ συχνά τα μέλη της Επιτροπής λένε ναι, ίσως να υπάρξουν απώλειες για το βόλιο κρέας σε αυτή τη συμφωνία, αλλά ό,τι χάσουμε στο βόλιο θα το ε, αποζημιώσουμε στο γαλακτοκομικό τομέα. Και χαίρομαι λοιπόν τώρα που σε αυτή τη συμφωνία για τη Νέα Ζηλανδία ε, συζητούμε τα θέματα αυτά, διότι θα καταστεί σαφές ε, πλέον στους γεωργού σε όλη την Ευρώπη ότι πρώτον και κυριότερον ό,τι χάνεται στο βόλιο κρέος, στη DTIP και στη ΣΥΤΑ και στο Μερκοσούρ, δεν ε, θα αποζημιωθεί μέσω κερδών στο γαλακτοκομικό τομέα οπουδήποτε αλλού. Και ό,τι χάνεται στο Βόρειο κρέα σε αυτές συμφωνίε ε, τελικά ε, θα ε, είναι ασήμαντο αν δούμε τι απειλέ αντιμετωπίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί, αν δούνε πόσο φιλόδοξε είναι αυτέ οι αποκαλούμενε συμφωνίε με τη Νέα Ζηλανδία. Για να μην αναφέρω δε για τι γίνεται με το αρνήσιο κρέα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα στην συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία που θα πρέπει να ε, προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς ως Επιτροπή Γεωργία. Θα πρέπει να ζητήσουμε αποκλεισμό των ευάλωτων τομέων. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και το Brexit. Θεωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα παράδοξο να υπάρξει γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργίας χωρίς να μην υπάρχει καν μία στο Brexit ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις τεράστιες απειλές ε, που προκύπτουν για τον Brexit, λόγω του Brexit για τους γεωργούς και στην Ιρλανδία αλλά και αλλού. Και αν λάβετε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία και να αγοραστούν 230.000 τόνους αρνιού και πρόβιου κρέατος από τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αγοράζει το 40% σημαίνει ότι θα δημιουργούν στρεβλώσεις εκτός και αν υπάρξει κάποιος μηχανισμός για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και πιστεύω ότι στην νομοδότησή μας θα πρέπει να ζητήσουμε αποκλεισμό οποιασδήποτε πρότασης ότι οι επενδύσεις που αποτελούν και το επίκεντρο αυτών των συμφωνιών ε, θα πρέπει να βρίσκονται εδώ. Θα πρέπει να ζητούμε να αποκλείονται αυτά τα προϊόντα από αυτές τις συμφωνίες, γιατί αυτές οι συμφωνίες θέλουν να βοηθήσουν τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και αυτό το οποίο βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο είναι ότι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις πολυεθνικές ε, και τους ε, γεωργούς που... Ε, έχουν μικρή παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλες πλέον. Είναι όλο και περισσότερες οι αντιθέσεις και το θέμα είναι ότι εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιανού το μέρος είμαστε. Ο κύριο Κάρθη είναι ο πρώτο που έλαβε το λόγο και δεν τον περιόρισα, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαι πιο αυστηρό γιατί στις 11.30 πρέπει να αρχίσει η συνεδρία των συντονιστών, οπότε α μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια σχόλια γιατί υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, οπότε σε αποφύγουμε τις επαναλήψεις. 1,5 λεπτό λοιπόν στους υπόλοιπους ε, ομιλητές, μου παρακαλώ. Ο κύριος Φλαζό. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως δεν χρειάζεται κανείς να μακρηγορήσει ε, για να πει ότι προκαλεί αυτή ε, η συμφωνία αυτοκτονική για τους παραγωγούς μας. Πρόκειται ουσιαστικά για εξαγωγή πρόβειου κρέατος, ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εγκληματικό αυτό, απλούστατα. Η πολιτική στρατηγική αυτή είναι εις βάρος των προβατοτρόφων που έτσι κι αλλιώς πνίγονται. Τι συζήτηση να κάνεις, δεν χρειάζεται μεγάλη συζήτηση εδώ, όπως και στη συμφωνία με την Αυστραλία. Θα πρέπει οπωσδήποτε το πρόβιο κρέα, αλλά και όλη η Γεωργία να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Αλλιώ. Εκείνοι που θα υπογράψουν αυτή τη συμφωνία θα είναι υπόλογοι ενώπιον των ε, κτηνοτρόφων. Όλο και περισσότερο πτωχεύουν και αυτοκτονούν οι κτηνοτρόφοι μας. Αυτά. Er Κύριε Σπαντακέτελα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συζήτηση είπαμε πολλά. Το κείμενο του κυρίου Νίκολσον αποτελεί καλή βάση για τη συζήτηση για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Νέα Ζηλονδία. Χαίρομαι ε, που μιλάτε για φιλοδοξία ε, στο εμπόριο. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν πολλοί κλάδοι της οικονομίας ε, και μετά το ρωσικό εμπάργο ο κόσμος ζητάει να κάνουμε συμφωνίες εξαγωγών. Ας πούμε, ε, η παραγωγή χειρίου κρέατος, αλλά και άλλοι τομείς. Δεν θα πρέπει βεβαίως να εθελοτυφλούμε, ε, να απαραγνωρίζουμε ε, τους ευαίσθητους τομείς. Θα πρέπει να διατρανώσουμε ως Επιτροπή Γεωργίας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου τη γνώμη μας. Χρειάζεται πολύ βαθιά ανάλυση και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη το Brexit. Προσωπικά δεν τρελαίνομαι για κρέας, ούτε πρόβιο, ούτε αρνίσιο. Αλλά εντάξει, δεν να κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η Γεωργία ε, ε, ε, θα πρέπει να παραγωνιστεί στη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών και στις διαπραγματεύσεις. Όχι, θα πρέπει να είναι ουσιαστικό τομέας μαζί με τους άλλους. Ευχαριστώ. Το πρόβιο κρέας είναι πολύ υγιεινό και το αρνίσιο το ίδιο. Το συνιστώ. Κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα συζητήσαμε προηγουμένως για την κλιματική αλλαγή και το νόημα όλων αυτών ε, των ταξιδιών των γεωργικών προϊόντων ανά την Ιφίλιο. Αλλά κύριε Νίκολσον, ε, θέσετε ένα ερώτημα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρωτήσατε πόσες συμφωνίες αντέχουμε ακόμα πριν καταρρεύσουμε τελείως και πριν κορεστούν απολύτω οι αγορέ μας. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται στο γάλα. Μας λένε τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν απελευθερώσουμε στα γαλακτοκομικά θα ε, έρθουν εισαγωγέ 450 με 800 εκατομμύρια. Γιατί η αγορά γαλακτός δεν είναι κορεσμένη. Από το 2015 μέχρι το 2016 στη Γερμανία από το Νοέμβριο σε ε, Νοέμβριο, χάσαμε πάνω από 4.000 γαλακτοκομικές επιχειρήσεις, 300 τη μέρα κλείνουν. Οι αγρότες πνίγονται ακόμα, δεν έχουν ανακάμψει από την κρίση αυτή. Και τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία για να έχουμε επιπλέον πίεση. Κατά τα άλλα, οι 18 ε, ε, λεπτά το λίτρο παίρνουν οι γαλακτοπαραγωγοί ε, στη Νέα Ζηλανδία, ούτε αυτοί μπορούν να ζήσουν από αυτές τις τιμές. και κάτι για τον προστατευτισμό. Ο προστατευτισμός δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Προστατευτισμός σημαίνει προστασία. Ο προστατευτισμός είναι πρόβλημα όταν είσαι εσύ υπεθετικός σε άλλες αγορές για να ξεφορτωθείς τα πλεονάσματά σου και από την άλλη να κλείσει την αγορά σου και να κατεβάζει τα ρολά και να κλείσει τα σύνορα για τα προϊόντα των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι η προστασία. Θα πρέπει πάντα να βλέπουμε ε, τι είναι σκόπιμο, τι είναι απαραίτητο σε εμπορικέ συμφωνίε και θα κάνουμε και τι τροπολογίε. Παρακαλώ. Ας ακούσουμε την έκκληση κυρία Χόιμπουχ ε, για να μην επαναλαμβάνουμε σχόλια που ήδη έχουν γίνει. Έτσι θα περιορίσουμε τη συζήτηση. Είναι ενδιαφέρον το θέμα της κατάστασης της γαλακτοκομικής αγοράς και της, του γάλακτος στην Ευρώπη. Κυρία Μίλλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή μας για τις σαφείς προτάσεις και τα σταρά τα λόγια του. Πραγματικά πρέπει να ληφθεί υπόψη η Γεωργία. Η Νέα Ζηλανδία βέβαια είναι άλλη τάξη μεγέθους από την Αυστραλία και άλλο δυναμικό ένα γαλακτοκομικό εργοστάσιο ε, μονοπολεί στην αγορά. Και εκτός του γάλακτος έχουμε και το αίγιο ε, και το πρόβιο κρέας. Και εδώ ασκούμε την κριτική μας, ε, επικρίνουμε την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Θέλουμε περισσότερη προφόρηση, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη συμμετοχή ως Επιτροπή Γεωργίας στις διαπραγματεύσεις. Και θα πρέπει να σκεφτούμε λογικές ποσοστώσεις και να τις απαιτήσουμε. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου φυσικά εδώ έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Η Γεωργία είναι μόλις το 10% του εμπορίου, προφανώς το ξέρουμε και εμείς αυτό, αλλά ακριβώς στην Επιτροπή Γεωργίας μας ενδιαφέρει η Γεωργία. Και έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για μας. Είναι και σημαντικός εργοδότης και εξασφαλίζει σημαντικές θέσεις απασχόλησης και η Γεωργία, όχι μόνο η βιομηχανία καλέ θέσει εργασία στη βιομηχανία, αλλά εμεί στη γεωργία πρέπει να σκεφτόμαστε και να προστατεύουμε. Με μια καλή συμφωνία ισορροπημένη και καλέ διαπραγματεύσει, νομίζω υπάρχουν ευκαιρίε με λίγη καλή θέληση. Δεν είμαστε κατά του ελευθέρου εμπορίου. Θέλουμε καλέ συμφωνίε. Σε ε, περίπτωση που υπογράψουμε τέτοια συμφωνία, είναι τουλάχιστον καλή. Η κυρία Ντελέ, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νίκολσον για το σχέδιο γνωμοδότησή του και να πω ότι κατά τη γνώμη μου η γνωμοδότηση του δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των Ευρωπαίων Γεωργών. Όπως και για τη συμφωνία με την Αυστραλία, θεωρώ και πάλι ότι τα ευαίσθητα προϊόντα όπως είναι ο γαλακτοκομικός καλάδος, το βόλιο και πρόβιο κρέας, θα πρέπει να ξερούνται από τις διαπραγματεύσεις. Κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνα με τον κύριο Κλάρκ, το διευθυντή της, Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής της Γεωργίας. Εγώ Πάντω, πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτού του κλάδου απέναντι σε πολύ ανταγωνιστικέ ε, αγορέ. Ελάχιστε είναι προοπτικέ και το ε, ενδιαφέρον τέτοιων συμφωνιών για, τέτοιους, ε, για τέτοιες αγορές. Είναι 4 εκατομμύρια μόνο οι καταναλωτές οι ενδιαφερόμενοι στους αντίποδες της Ευρώπης. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης στην έκθεση είναι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Ο κύριος Τωραμπέλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κάποια στοιχεία πρώτα η Νέα Ζηλανδία έχει περισσότερες γαλακτοφόρες αγελάδες από ό,τι κατοίκους. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε ε, ε, μία γαλακτοφόρα αγελάδα για 21 κατοίκους. Επίσης, 88% ε, του γάλακτος το εξάγει η Νέα Ζηλανδία. Εμείς το 14% μόνο το εξάγουμε και είναι φυσικό γιατί θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στην γαλακτοκομική παραγωγή και δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτό τον ευρωπαϊκό κλάδο. Όπως ε, και ο Καναδάς στις ε, διαπραγματεύσεις της ε, ΣΕΤΑ, ο Καναδάς προστάτευσε την γαλακτοκομική αγορά. Είναι η πιο ρυθμισμένη αγορά και στην, στον κόσμο με τις μεγαλύτερες αμοιβέ για τους κτηνοτρόφους, τους γαλακτοπαραγωγούς και την προστάτευσε. Δεν είναι βρισιά η προσβολή που θέλουμε να προστατεύσουμε τους παραγωγούς μας. Και επίση το Brexit, το είπα και προηγουμένω όταν το 1973 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε παραχωρήσει πολύ ευνοϊκέ για το πρόβιο κρέα ε, τη Νέα Ζηλανδία με πραγματικά πολύ χαμηλού ε, δασμού ε, που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Μετά το Brexit θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτές τις συμφωνίες, γιατί θα βγει από το, την Ευρωπαϊκή Ένωση το Brexit ή είναι κεκτημένο αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δώσαμε στη Νέα Ζηλανδία με την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει με τον Brexit. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν σχετικά και οι σχετικές ε, διατάξεις στη συμφωνία με τη Ζηλανδία, με την Νέα Ζηλανδία. Κύριε Ταραμπέλα, μπορείτε να πιείτε ένα καφεδάκι μαζί με τον κύριο Νταντέν και τον ε, ε, κύριο Μπαρνιέ που είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και να του επισημάνετε όλα αυτά τα θέματα για τον Brexit και τη Γεωργία. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στην προηγούμενη συζήτηση ε, για τις εμπορικές συμφωνίες, ο Τζον Κλάρκ μίλησε για σχετική συμπληρωματικότητα. Καλή τύχη στους διερμηνείς. Απαντώντας στα δικά μου σχόλια και σχόλια άλλων, όπου θα βλέπαμε μια κατάσταση όπου θα είχαμε τα ίδια αγαθά, να διασταυρώνονται το βράδυ στα πλοία. Και μου είπαν, όχι θα υπάρχει λέει μια σχετική συμπληρωματικότητα, αυτό είπε ο κύριος Κλάρκ. Και μάλιστα παράδειγμα ακούσαμε και για τα αμύγδαλα. Ε, πώς θα παράγει η Ευρώπη, θα εισάγει αμύγδαλα. Ποια είναι η συμπληρωματικότητα. Εμείς τι θα εξάγουμε σε τέτοιες μεγάλες ποσότητες που θα διασταυρώνεται με ένα μεγάλο πλοίο από την άλλη πλευρά. Πού είναι η σχετική συμπληρωματικότητα. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, το Σάββατο ε, μίλησα με ένα Γιωργό από το Δυτικό Ντάραμ ε, που έχει ε, πρόβατα και βοηδή και κάτι που δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση μέχρι τώρα και μου επισήμανε είναι το θέμα της ευζοίας, της καλής μεταχείρισης των ζώων. Στην Νέα Ζηλανδία έχουμε πολύ μεγαλύτερα κοπάδια και τα αρνιά μένουν στα ε, στους ε, λόφους, δεν ξεχυμάζουν και γι' αυτό έχουμε μεγάλη χρησιμότητα των αγέννητων αμνών και των προβάτων. Και μάλιστα οι συνθήκες ε, θανάτου δεν είναι και πολύ ευχάριστες. Είναι επώδυνη διαδικασία και ο επώδυνος πολλές φορές ο τοκετός γιατί δεν υπάρχει βοήθεια από κτηνοτρόφο, από το κτηνίατρο, συγγνώμη. Οπότε είναι πολύ ε, αρνητική η διάκριση βάρος των Ευρωπαίων γεωργών που τηρούν και κτηνοτρόφων που τηρούν πολύ υψηλότερες προδιαγραφές καλής μεταχείρισης των ζώων. Και σε ό,τι αφορά το Brexit, σίγουρα οι εμπορικές συμφωνίες είναι εξορισμού και εκφύσεως περίπλοκες και το Brexit θα είναι ε, περίπλοκο και μάλιστα ο συνδυασμός με τις εμπορικές συμφωνίες το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο και περίπλοκο και ένα από τα πιθανά ζητήματα που θα ανακύψουν είναι το ότι η ε, Βρετανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει απεγνωσμένα να συνάψει κάποιε εμπορικέ συμφωνίε με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία σίγουρα ε, είναι χώρε στόχο γιατί μιλούμε την ίδια γλώσσα, έχουμε κοινού δεσμού και ούτω καθεξή. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία θα είναι σε πολύ καλή διαπραγματευτική θέση για να έχουν σκληρές διαπραγματεύσεις και να πετύχουν παραχωρήσει από το ΕΒ που θα είναι απεγνωσμένο να συνάψει τέτοιες συμφωνίες. Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι θα κατακλειστεί το ΕΒ με φθηνό αρνήσιο και πρόβιο κρέας. Και ε, μετά την επεξεργασία το κρέας ε, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πια και η χνηλασιμότητα περιπλέκεται τι θα γίνει. Θα έχουμε ξεχωριστό σύστημα ε, δασμολογικών ποσοστώσεων ε, ή δασμών όπου ε, το κρέας, το κατεργασμένο θα υφίσταται σε διαφορετικές, θα υπόκειται σε διαφορετικούς δασμούς αν είναι του, Ευρω... του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε και σε άλλους πιο υψηλούς όταν προέρχεται από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, πώς θα γίνει η χνηλασιμότητα όταν μιλούμε για αλεσμένο κρέας, για κοιμά, για καταργασμένο κρέας. Θα είναι πολύ δύσκολο και για τους Βρετανούς γεωργούς φυσικά κάτι τέτοιο. Πώς να πούν όχι στην εισαγωγή φθηνού κρέατος από Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Μερικοί καταναλωτές μόνο φθηνού κρέας μπορούν να, να αγοράσουν και δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι αδιαφορούμε και για αυτούς. Ευχαριστώ. Επειδή εσεί δεν είχατε λάβει το λόγο στην προηγούμενη συζήτηση για την Αυστραλία, σα επέτρεψα να μακρηγορήσετε κάπω. Κυρία Νόιχ, ο κύριο Σνέκοφ, συγγνώμη, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, κύριε Κλάρκ, συμφωνώ με τη, τη γενική κατεύθυνση και τα βασικά σημεία της γνωμοδότησης Νίκολσον Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε κάποιους παραγράφους γιατί η οικονομία της Νέας Ζηλανδίας είναι πολύ πιο φιλελεύθερη και έχει μεγαλύτερο εξαγωγικό προσανατολισμό από την ευρωπαϊκή. Πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές προανέφεραν ήδη τους ευαίσθητους τομείς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως στο εγωπρόβιο κρέας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο πληθυσμός ε, της Νέας ε, Ζηλανδίας είναι μόνο 4,7 εκατομμύρια. Εισάγει όμως, ε, εξάγει όμως η χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεωργικά προϊόντα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει γεωργικά αγαθά προς τη Νέα Ζηλανδία 450 εκατομμύριων μόλις ε, ευρώ. Δηλαδή ε, τέσσερις φορές ε, λιγότερος όγκος ε, από την Ευρώπη προς τη Νέα Ζηλανδία. Επίσης η παραγωγή μελιού στη Νέα Ζηλανδία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι το μελισσοκέρι και το μέλι θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εμπορική συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε, στις γεωγραφικές ενδείξεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και με τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν επιχειρήματα βέβαια κάποιων χωρών μελών για τα γενώσιμα προϊόντα. Άρθρα 22, 23 και 24 από τη Συμφωνία TRIPS. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πολύ σημαντικές ε, για τη γαστρονομική μας κληρονομιά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων μας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Επίσης πιστεύω ότι η Νέα Ζηλανδία θα πρέπει επίσης να επιδιώξει να αναγνωριστούν από την Ευρώπη οι δικοί της κανόνες. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τον Brexit. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Για το πρόβιο και βόηο κρέας, το 40% των εισαγωγών από τη Νέα Ζηλανδία κατευθύνεται ε, προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή, ε, αυτό το στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ένα νομικό κενό που ίσως ε, φέρει σε δύσκολη θέση και ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους ακτινοτρόφους και παραγωγούς. Θα καταθέσω τροπολογία στη γνωμοδότηση του κυρίου Νίκολσον. Ελπίζω να προλάβαμε στην προθεσμία και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με το συντάκτη γνωμοδότησης. Η κυρία για ένα λεπτό. Η μόνη διαφορά που θα μπορούσα να ε, διαπιστώσω σε σχέση με τη Νέα Ζηλανδία είναι ότι υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλες εξαγωγές και πιστεύω ότι εδώ θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να απαιτήσουμε ε, επίπεδα ευρωπαϊκών προτύπων και σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο όπως ε, πολύ σωστά ακούστηκε από τον συνάδελφο Μπλάνινγκ σε θέματα ευημερία των ζώων, θα πρέπει να συγκρίνουμε τα πρότυπα και σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, τροπολογίες. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει τροπολογία εδώ, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό εάν μπορεί να επηρεάσει τη συζήτηση να τεθεί στην Επιτροπή Ίντα όταν θα συζητηθούν τα θέματα αυτά στην ε, αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Κλάρκ, παρακαλώ. Thank you, I'll, not repeat anything I've said. Δεν θα επαναλάβω όσα σας είπα και προηγουμένως. Ε, τέσσερα πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, συμφωνούμε απολύτως ε, με την ουσία της γνωμοδότησης, την έκκληση για ισορροπία, την ανάγκη να διατηρήσουμε ευαίσθητου τομεί, ε, και όπως και στην περίπτωση της Αυστραλίας ε, πλήρη αποκλεισμό όλων των ευαίσθητων τομέων δεν είναι ρεαλιστικό για δύο λόγους. Πρώτον, ε, γιατί ο διαπραγματευτικός εταίρος ποτέ δεν θα δεχθεί να αποκλειστούν όλου τους τομεί που του ενδιαφέρουν ω εξαγωγή. Δεν είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση. Και δεύτερον, διότι είτε σα αρέσει είτε όχι, οι κανόνες του ΠΟΕ προβλέπουν ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να καλύπτουν ουσιαστικά όλο το εμπόριο, το 90% όλου του εμπορίου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε λοιπόν τη γεωργία εξ ολοκλήρου και να περάσουμε τις δοκιμέ ε, του ΠΟΕ. Σίγουρα υπάρχουν βεβαίω εναλλακτικέ λύσεις αντί του πλήρου αποκλεισμού. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι πόσες ε, ε, συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών μπορούμε να διαπραγματευτούμε μέχρι να φτάσουμε στο όριο όσον αφορά το βόλιο, το αρνήσιο κρέα κλπ. Το θέμα δεν είναι πόσε συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών, αλλά πόσο είναι ο σιωρευτικό όγκο που μπορούμε να εισάγουμε συνολικά από όλε αυτέ τι συμφωνίε. Και έχει γίνει μια αξιολόγηση ε, τη σιωρευτική ε, επίδραση ε, και για συμφωνίε οι οποίε συνέφθηκαν προσφάτω και για αυτέ οι οποίε είναι εν εξελίξη. Ουκρανία, Βιετνάμ, Νότιο Αφρική. Και φυσικά προσβλέπουμε και στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Τίτυπ, τη Μερκοσούρ, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό και τη Χιλή. Έγιναν αυτά και πριν από κάποιους μήνες δημοσιεύτηκε και η έκθεση και επίσης θα γίνει και μια αξιολόγηση επιπτώσεων για τη συμφωνία και της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας ξεχωριστά, όταν θα έχουν εγκριθεί και εντολέ από πλευρά Συμβουλίου για το φθινόπωρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, θα κάνει διεξοδικότατε αξιολογήσει επιπτώσεων όλων αυτών των συμφωνιών, που θα περιλαμβάνει φυσικά και το γεωργικό τομέα, ο οποίο θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των δύο διαπραγματεύσεων. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Ταραμπέλα ρώτησε για το Brexit και τη μοίρα των ποσοστώσεων του ΠΟΕ για ε, το πρόβιο και το αρνήσιο κρέας. Ε, πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα ήταν χρήσιμο να αναφέρει το Brexit, ε, όπως έγινε και στη γνωμοδότηση με την Αυστραλία. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σχέση αυτό. Και να απαντήσω και στον κύριο Ταραμπέλα ότι ναι, εξετάζουμε το μέλλον ε, αυτού της ε, ρήτρα του ΠΟΕ, διότι όπως είπατε και εσείς, το Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνει περίπου το 40% του πρόβειου κρόατος που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουμε υπόψη και σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σνίκολσον. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κλάρκ για την απάντηση. Όλοι σεβόμαστε τις απόψεις του και είναι και πολύ σαφής. Μήπως η γραμματεία θα μπορούσε να έχει ε, αντίγραφα τη έκθεση αυτή τη μελέτης αντικτύπου που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας τα μοιράσει γιατί θα είναι καλό ανάγνωσμα και ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγέ πρόβειου και βοηού κρέατο, ότι θα καταρρεύσει η αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστρεψε η ίδια τον κλάδο αυτό, ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δίνει τις ενισχύσεις. Όταν έκανε την ενίσχυση στρεματική αντί ε, να είναι αναζώο, κατέστρεψε παντού στην Ευρώπη όλο τον κλάδο του βοηού και του προβίου κρέατος. Αν θέλεις να έχεις δοτροφία και προβατοτροφία, θα πρέπει να επιστρέψεις στις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις και στο γαλακτοκομικό. Γιατί αν έχουμε στραφεί στην παραγωγή ε, γαλακτός δεν θα έχουμε την παραγωγή κρέατος που χρειαζόμαστε. Συγγνώμη, αλλά είναι το αγαπημένο μου θέμα. Εμείς αυτό καταστρεφόμαστε, δεν χρειαζόμαστε τις ε, εισαγωγέ για να καταστραφούμε από τη Νέα Ζηλανδία. Έχουν το πλεονέκτημα της οικονομίας κλίμακος και ο κύριος Ντές αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από εμά. Αλλά, συνάδελφοι, εμείς κάνουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή διεθνούς εμπορίου, αν είναι προστατευτική η γνωμοδότησή μας, δεν θα τη λάβουν καν υπόψη στην ίντα. Θα πρέπει να τους υποβάλουμε μια γνωμοδότηση που θα την συζητήσουν, που θα την εντάξουν στην έκθεσή τους και θα τη σεβαστούν για να μπορέσουμε εμείς από εκεί και πέρα να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή αυτή. Σημειώνω αυτά που είπε ο κύριος Κλάρκ και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να τα συμπεριλάβω και στη νομοδοτήση. Είπα και προηγουμένω πόσο λίγο χρόνο είχαμε με τον κύριο Αντρέο για τι νομοδοτήσει μα. Ιδιαίτερα αυτά που είπατε για την ευημερία των ζώων και τη βιωσιμότητα και την αηφορία. Πολύ σημαντικά. Και για το Brexit, βεβαίως πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό και να το συμπεριλάβουμε, αλλά εγώ πώς το βλέπω στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν. θα γίνουν διαπραγματεύσεις και για τις ίδιες τις ποσοστώσεις. Και δεν φανταζομαι ότι θα υπάρξουν άλλες χώρες που θα θέλουν να αναλάβουν το βάρος των προβλημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και να το απαλλάξουν από τα προβλήματα. Θα τα δούμε αυτά τα θέματα που συνδέονται με τον Brexit, δεν είναι του παρόντος. Και ο κύριος Άντρο, εγώ θα συνεργαστούμε για να έχουμε αντίστοιχη θέση και προσανατολισμός προς τον Brexit. Προσβλέπω συνεργασία και με τους σκιώδες ηγητές για να έχουμε ενιαία θέση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά και πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει οπωσδήποτε εμεί στη Γεωργία να έχουμε λόγο για τις εμπορικέ αυτές διαπραγματεύσεις. Γιατί για πολύ καιρό μας είχαν παραγωνίσει, για να μην πω ότι είχαμε αυτό παραγωνιστεί. Έχει έρθει η ώρα να ακουστεί η φωνή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέχρι την πρώτη σε, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, 11 το μεσημέρι, έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες. Ε, συμφωνώ με την θέση που εκφράσατε ε, για το και το παράπονο για το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, αλλά αν θέλαμε να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μας από την Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου, ήμασταν υποχρεωμένοι να προβλέψουμε τέτοιο στενό χρονοδιάγραμμα. Και επίσης είναι τόσο φιλελεύθερη θέση τη. Ε, διεθνούς, ε, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου που αν δεν προλαβαίναμε να υποβάλουμε την ε, έκθεση, την γνωμότατησή μας δεν θα ακουγόταν καθόλου θέση του Γεωργίου. Και από τον Επιτροπο και από την κυρία Βάλστρομ είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις ε, θα συνεχίσουμε να πετούμε μεγαλύτερη ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα γεωργικά θέματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δίνουμε τα γεωρικά ζητήματα ως αντάλλαγμα για πλεονεκτήματα που διεκδικούμε σε άλλους τομείς, υπηρεσίες, οικονομικά, χρηματοοικονομικά και το καθεξής. Αλλά μερικές φορές ε, είναι η γεωργία το αντάλλαγμα που δίνουμε, το ανταλλακτικό νόμισμα. Θα πρέπει να γίνονται ε, μελέτες επιπτώσεων και αντικτύπου για όλες τις πλευρές ε, για να γνωρίζουμε πώς θα επηρεάσουν οι διαπραγματεύσεις. Και επίσης θα ήθελα να καλέσω τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ να στηριχθούν ε, και στην πραγματικότητα, να λάβουν υπόψη την πραγματικότητα και την κατάσταση των Ευρωπαίων Γεωργών. Θερμή έκκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ θερμά τους ηγητές, τους συντάκτες γνωμοδότης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του συναδέλφους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Τρίλεπτη διακοπή και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίε των συντονιστών. Η υπόλοιπη επιτροπή θα συνεχίσει τη δημόσια της συνεδρίασης στις 3.